Okay. Welcome to everybody. We can start now. Καλώς ορίσατε όλοι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αν έχετε την καλοσύνη καθίστε. And so we have uh, different items, very interesting. Έχουμε διάφορα σημεία προσυζήτηση, μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση και στο τέλος θα έχουμε μια ενημέρωση από την ε, DG Cult ε, για το follow-up του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Δίνω το λόγο στον πρώτο εισηγητή Μισελ Ρεϊμόν για το σημείο 12, επιδίωξη ανανεωμένη συνένεση όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητική ιδιοκτησία στην εσωτερική αγορά, σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αρμόδια τη ουσία επιτροπή είναι η Γιούρη. Ας ακούσουμε τώρα την παρουσίαση. Δίνω το λόγο στον κύριο εισηγητή. Συνεχίζουμε συνεχίζω στα τελικά εγώ μετά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρώτο σχέδιο έχει σταλεί στους Σκιώδης, από γνωρίζω χθες ή προχθές. Προτείνω πέντε σημεία σε αυτό το σχέδιο το πρώτο είναι ότι στόχος κλειδί ενός σχεδίου δράσης πρέπει να είναι η εργασία με αξιόπιστα δεδομένα. Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται και παρέχονται από τον ε, σχετικό τομέα, από τη βιομηχανία που ε, φυσικά ενδιαφέρεται ε, ο κλάδος αυτός να αντιμετωπίσει την κατάχρηση τη διανοητική ιδιοκτησία. Χρειαζόμαστε λοιπόν αντικειμενικά στοιχεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα αποκτέουμε και να τα επεξεργαζόμαστε. Το Γραφείο Εναρμόνισης και Εσωτερικής Αγοράς θα πρέπει να επιφορτιστεί με το καθήκον να παράσχει αυτά τα στοιχεία. Ε, το δεύτερο και το τρίτο σημείο ε, πάνε μαζί. για την καινοτομία και τη δημιουργικότητα θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε όλες οι πληροφορίες για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας να είναι ως το δυνατόν πιο διαφανείς. Αυτό συνάδει με τη νέα νομοθεσία περί copyright που συζητείται στην Γιούρη και που θα συζητηθεί με στους επόμενους μήνες για να έχουμε μια καινοτόμο νέα νομοθεσία περί copyright θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι εύχρηστη. Δηλαδή θα πρέπει ο κόσμος να μπορεί να γνωρίζει πότε ισχύει και πότε όχι, πρέπει οι προφορές να είναι διαφανείς, πότε επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και πότε όχι ε, αυτή η νομοθεσία και πότε ισχύουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και πότε όχι για ένα συγκεκριμένο στοιχείο. Αυτά είναι τα σημεία 2 και 3. Να τονίσω επίσης ότι η ανοιχτή πρόσβαση στις πληροφορίες, η ανοιχτή γνώση, η ανοιχτή πρόσβαση ενδεχομένω και στη γενετική ιδιοκτησία είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ε, ανάπτυξή μας ε, εφόσον η ενιαία ψηφιακή αγορά αποτελεί ζήτημα κλειδί για την επόμενη πενταετία για την Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για το Κοινοβούλιο όσο και για την Κομισιόν είναι σημαντικό αυτό το σημείο για την επιβολή λοιπόν των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ε, πρέπει να πούμε ότι δεν μας συμφέρει η ελέγχη να είναι όσο το δυνατόν αυστηρότερη. Θέλουμε να ε, βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την ανοιχτή έρευνα και την ανοιχτή γνώση. Το πέμπτο σημείο είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. Τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Φυσικά οι απομιμήσεις προϊόντων ε, δεν παραβιάζουν απλά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά είναι και επισφαλή και μπορεί να βλάψουν την υγεία. Ε, δεν θέλω να συνδυάσουμε μαζί αυτά τα δύο ζητήματα, θέλω να τα εξετάσουμε ξεχωριστά, διότι χρειάζονται και τα δύο μια πιο σοβαρή προσέγγιση. Αυτό αναφέρω στο πέμπτο σημείο. Αυτά κατά βάση. Με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ε, Ευχαριστούμε κύριε Ρέμο. Έχουμε ήδη μια αίτηση από τον συνάδελφο Ζουλό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο και μπορείτε να εγγραφείτε για να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά του και τις πληροφορίες που παρέχει στη γνωμοδότησή του. Η παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη ο οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων. Φυσικά όλοι συμμεριζόμαστε τη βούληση να αυξήσουμε τη διαφάνεια και να βασίσουμε οποιαδήποτε δράση καταπολέμησης των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε αξιόπιστα δεδομένα. Πολλέ μπορεί να είναι οι αντιδράσει μας σε αυτά τα προβλήματα. Εξήγησε διάφορα ζητήματα ο κύριος Ρέιμον. Μπορούμε να βρούμε κι άλλα, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κάποιο περιορισμό για το μέγεθος της αρχικής γνωμοδότηση. Να σα δώσω δύο παραδείγματα. Το πρώτο αφορά το ζήτημα των κερδών που αποκομίζουν ε, οι πλατφόρμες φιλοξενίας και που χρησιμοποιούνται για το παράνομο κατέβασμα αρχείων και το δεύτερο είναι η ε, παραποίηση κατά την πώληση online έργων τέχνης. Όσον αφορά τις πλατφόρμες φιλοξενίας, ε, αυτές βασίζονται στον εξής απλό συνδυασμό της διαφήμισης και της συνδρομής των χρηστών οι οποίοι με τη συνδρομή μπορεί με αυτόν τον τρόπο, πληρώνοντα μια συνδρομή, να κατεβάζουν τα αρχεία πιο γρήγορα και να έχουν περισσότερο χώρο αποθήκευση. Οι ιστοσελίδε αυτέ ε, που αποτελούν ε, βάση για ένα κομμάτι τη ροή παράνομων αρχείων ουσιαστικά αποκομίζουν κέρδη από τις παραβιάσεις στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Το δεύτερο παράδειγμα παρότι σχετίζεται με τον ψηφιακό κόσμο, είναι η όλο ένα και μεγαλύτερη αύξηση των παραποιημένων εργών τέχνης, των πλαστών εργών τέχνης που κυκλοφορούν στην αγορά χάρη στην ανάπτυξη των online πωλήσεων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται, δεν δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της αυθεντικότητας των έργων αυτών, οπότε ο κόσμος μπορεί να ε, αγοράσει κατά λάθο ε, πλαστά έργα τέχνης τα οποία κυκλοφορεί μετά στην αγορά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, και οι τροπολογίες που θα προταθούν ε, σίγουρα θα αναφερθούν και σε περισσότερους τομείς από τα παραδείγματα που αναφέρω εγώ. Απλά έχω να πω ότι πολλές διαφορετικές μπορεί να είναι οι απαντήσεις θα πρέπει να συνδυάζουν την ευαισθητοποίηση, τι συμφωνίε μεταξύ των διαφόρων κλάδων και σίγουρα και τις κυρώσεις και τη διαβούλευση με διάφορου φορείς ε, του κλάδου. Όλα αυτά είναι αναγκαία για να καταλήξουμε σε σύμφωνες και καλές πρακτικές για να καταπολεμήσουμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτά ήθελα να προσθέσω. Ευχαριστούμε τον ε, κύριο εισηγητή για την εργασία του. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Πέτρα Κάμερβερτ. Ευχαριστώ για εμάς ε, τις σοσιαλδημοκράτησες είναι σκιώδη ηγητής ο συνάδελφός μου Γραμματικάκης, ο οποίος όμως δυστυχώς κολλείεται σήμερα, αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για τον ε, ελληνικό προεκλογικό αγώνα. Έτσι μου έχει γράψει εδώ ορισμένα και μου ζήτησε να τα ε, παρουσιάσω. Ένα από τα κέρια θέματα κατά την άποψη του Γραμματικάκη θα πρέπει να είναι και η βελτίωση, η επιτάχυνση δηλαδή της απονομής δικαιοσύνης σε αστικές διαφορές. Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο. για τους δημιουργούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να προστατεύσουν αλλιώς τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει αυτό να ισχύει για όλες τις ε, σχετικές υποθέσεις και θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή από τα δικαστήρια να μην υπάρχουν και παραβιάσει θεμελιωδών δικαιωμάτων και αλλιώ να υπάρχει μια εύλογη ισορροπία όταν μιλούμε εδώ για το διαδίκτυο. Χρειάζονται επίσης συγκεκριμένες ενημερωτικές εκστρατείες, σύμφωνα με τον κύριο Γραμματικάκη, για να υπάρξει συνειδητοποίηση ιδίως από τις νεότερες γενναίες που μεγαλώνουν μέσα στην εποχή του διαδικτύου σχετικά με το τι σημαίνει διανοητική ιδιοκτησία και ότι επομένως οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να αμείβονται για την δημιουργικότητά τους. Πρέπει λοιπόν να αναπτυχθεί μια συνείδηση για την αξία των έργων του δημιουργού βασικός στόχος του σχεδίου δράσεως θα πρέπει να είναι εκτός από την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ελευθερίας και μια δημιουργία μιας ευρύτερης νομικής προσφοράς που θα παίξει ένα ρόλο κλειδί για την ανάπτυξη, για την δημιουργία απασχόλησης στους χώρους του πολιτισμού, καθώς και για την πολιτική, πολιτιστική συγγνώμη, ε, πολυφωνία. Ιδίως σε αυτή την περίοδο κρίσεως όπου έχει υποστεί βαριές τομές το, το δημιουργικό πολιτιστικό έργο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δίκαιη δηλαδή μεταχείριση των καλλιτεχνικών δημιουργών. Ασφαλώς και αυτό αποτελεί ένα στόχο του σχέδιου δράσεως. Σημαντικό λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ε, μια ευρύτερη προσφορά μέσων, ε, προσφυγών δηλαδή, στους δημιουργούς. Και βεβαίως και για να πληρώνονται οι δημιουργοί επιγραμμικά, online. Για την αμοιβή τους που καμιά φορά είναι 2,5 ευρώ το κομμάτι, είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτή. Είναι πολύ περίπλοκο. Και γι' αυτό καμιά φορά οι άνθρωποι παρετούνται και από την ε, πληρωμή. Πρέπει να γίνει προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή και να τονιστεί επίσης το γεγονός ότι παραποιημένα προϊόντα δεν σημαίνουν μοναχά μείωση του εισοδήματο των ε, σοβαρών δημιουργών, αλλά και σε απώλεια της θέσεων απασχόλησης, σε αύξηση κόστους προσφυγών κλπ. Και βεβαίως και σε ενίσχυση ενός μεγάλου τμήματος της οργανωμένης εγκληματικότητας. και βέβαια και στη μείωση της ασφάλειας καταναλωτών, ε, για παράδειγμα λόγω παραποιημένων φαρμάκων. Χρειάζονται λοιπόν προληπτικά μέτρα, χρειάζονται συστήματα καταγραφής για την καταγραφή δηλαδή των παραβιάσεων των δικαιωμάτων των δημιουργών και χωρίς βεβαίως να υπάρξει ε, παραβιάσεις, να υπάρξουν ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρέπει σε συνεργασία με τα άλλα θεσμικά όργανα, θεσμικά όργανα να αναζητηθούν τρόποι και για τη λήψη συγκεκριμένων νομοθετικών μέτρων. Αυτά τα έχει πει ήδη ο Επίτροπος Oettinger, έχει ανακοινώσει ο Επίτροπος Oettinger, ότι δηλαδή μπορούν να αναμένουμε σχετικές προτάσεις ήδη φέτος, τις οποίες όλοι και όλες αναμένουμε βεβαίως με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτά που διάβασα είναι ορισμένες συστάσεις δικές μας, ή πάντως ε, του κυρίου Γραμματικάκη, για συμπληρώσεις στο κείμενο της εκθέσεως. Ευχαριστούμε Πέτρα. Κριστίνα Λιμπάσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή με τη σειρά μου για την ξεκάθαρη παρουσίαση του θέματος. Μια ερώτηση για την παράγραφο 4. Γιατί εκεί αναφερθήκατε στην πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στα πορίσματα επιστημονικών εργασιών. Να μην λησμονούμε όμως ότι τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας λαμβάνουν χαρακτήρα εμπορικό. Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά και όλο και εντονότερα. Καμιά φορά γίνονται και αντικείμενο εμπορικών διαπραγματεύσεων και βεβαίως και εμπορικών ευρεσιτεχνιών. Τρίτον, πρέπει πράγματι να σεβόμαστε τα δικαιώματα ε, διανοητικής ιδιοκτησίας. Πώς θα συμφιλιώσετε τότε λοιπόν αυτό που ζητάτε, την πρόσβαση δηλαδή μέσω διαδικτύου επιγραμμικά στα απορίσματα της επιστημονικής έρευνας και στην ανάγκη προστασίας τους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως, λέει κυρία Μακάρτιν, πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αν θέλουμε να είμαστε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό και βεβαίως όταν ε, θα έχουμε τα δικαιώματα αυτά πρέπει να επιβάλλεται η προστασία τους. Ερωτήσεις προς τον εισηγητή. Ιδίως στην παράγραφο 1 του σχέδιου του αυτά λέτε να μην βασίζονται μοναχά στα δεδομένα που προσφέρει η ίδια η βιομηχανία. Τι ακριβώς εννοείτε. Μπορούν να είναι άτομα, μπορούν να είναι εταιρείε, μπορούν να είναι επιχειρήσεις. Αυτοί όμως είναι, δηλαδή αυτοί που παράγουν το διανοητικό έργο, είναι αυτοί που, θεωρούν, που μπορούν μάλλον να εκτιμήσουν εάν υφίστανται παραβία στα δικαιώματά τους αυτά ή όχι. τι ακριβώς εννοείται. Δεύτερο. Παράγραφος 4 του κειμένου σας. Έρευνα και γνώση που αποκτάτε μέσω της έρευνας. Δεν νομίζω ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι αποκλειστικά. Μπορούν να συμβαδίζουν. Αν κάτι δηλαδή έχει μεγάλη αξία, εάν δεν προστατεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας, ε, αν δεν τυχάνουν προστασίας δηλαδή, δεν θα υπάρχει και το οικονομικό ενδιαφέρον για να γίνουν σχετικές επενδύσεις. Για την τελική σας παράγραφο, είναι λίγο ασαφές για μένα, σε ποιο είδους ασφάλεια της υγείας αναφέρεται ο εισηγητής. Θα ήθελα να υπάρξουν ορισμένα, θα ήθελα να αναφέρει μάλλον ορισμένα παραδείγματα για να διευκρινίσει το επιχείρημα της παράγραφου 5. Είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την προστασία των διανοητικών δικαιωμάτων και ιδίως για τους ερευνητές. Ευχαριστούμε ε, κύριε Στρογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Δύο είναι οι ερωτήσεις μου προς τον εισηγητή επί σειρά ετών επεξεργαζόμουν στατιστικά δεδομένα ε, στον τομέα του πολιτισμού και έχω κάποιες αμφιβολίες ως προς την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιούμε για την κατάρτιση εκθέσεων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση για τα δεδομένα τα οποία εσείς χρησιμοποιήσατε για να συντάξετε την έκθεσή σας. Δηλαδή πειρατεία, σε διάφορους τομείς, από μυς, παραδείς και τα λοιπά. Μπορούμε να πούμε σήμερα ότι τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι αξιόπιστα, είναι ικανοποιητικά, είναι δε και σωστά, αληθή. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι με βάση τα όσα γνωρίζουμε μπορούμε να συντάσουμε εκθέσεις που και αυτές θα είναι αξιόπιστες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Διακόνου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να πω το εξής. Βέβαια δεν πρόκειται τόσο για ερώτημα, αλλά για ένα σχόλιο προσωπικό. Με βάση την εμπειρία. Τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι το σημαντικό. Την πραγματικότητα πρέπει να γνωρίζουμε διότι εδώ κινούμαστε μέσα σε μια νομική περιοχή διαφοράς, ε, διαμάχης ε, δικαστικής. Θα ε, το εξηγήσω για να με καταλάβετε. Όταν μιλάμε για δικαιώματα δημιουργού, οι καλλιτέχνες φαίνεται να είναι το θύμα. των φορέων μετάλλευση ενός συστήματος και οι πολιτές ή οι μεσάζοντες είναι οι εχθροί εντό εισαγωγικών. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός. Στη Ρουμανία υπάρχει ένα ζήτημα με μια ταινία από τη δεκαετία του 70 επί Τσαουσέσκου δηλαδή Ένα μέρος της ε, ταινία χρησιμοποιήθηκε για να δημιουργηθεί ένα μικρής διάρκειας διαφημιστικό σποτ. Και υπάρχει μια δίκη τώρα πάνω σε αυτό το θέμα. Μου είχαν πει και όλα να συμμετάσχω σε αυτό το σποτ. Εγώ είπα όχι, δεν κάνω διαφημίσεις, δεν θέλω να συμμετέχω σε καμία διαφήμιση. Ιδίω εφόσον είχε γυριστεί επί Τσαουσέσκου η ταινία αρχικά. Υπάρχει λοιπόν τώρα καστική διαμάχη αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ. Δεν θα πρέπει η νομοθεσία να αφήνει παραθυράκια και για, να, και για καταχρήσεις ή παραβιάσεις των δικαιωμάτων δημιουργού. Για τη μουσική, για παράδειγμα. Οποιοδήποτε είδος. Συγκεκριμένα στη Ρουμανία πάλι έχουμε μια δικαστική διαμάχη με την όπερα του Βουκουρεστίου. γιατί στην ε, Εθνική Όπερα παίζονταν κάποιες κλασικές όπερες, αλλά δεν είχε στην προκειμένη περίπτωση, ήταν ε, όπερες του Μότσαρτ, δεν είχαν ε, καταβληθεί τα πνευματικά δικαιώματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν νομικά κενά εδώ. Είναι λεπτό το θέμα. Γενικότερα το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό γιατί δεν υπάρχει και κάποια συνθήκη, κάποιο νομοθέτημα που να είναι παρκώς αυστηρό και να ορίζει το πλαίσιο. Στην προκειμένη περίπτωση ένα δίκο βρίσκονταν οι καλλιτέχνες και δεν ήταν αυτοί τα θύματα. Πάντως το θέμα γενικά είναι σοβαρό. Στο διαδίκτυο τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, επικρατεί πολύ μεγάλη σύγχυση. Πάντω έχω εμπιστοσύνη στον εισηγητή και ελπίζω να έχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Διακονού. Πριν ε, δώσω το λόγο στον κύριο εισηγητή, να κάνω δύο ερωτήσει προσωπικέ. Κάτι πρώτα απ' όλα που θα θέλαμε να εμβαθύνουμε ενδεχομένω. Λέτε στο πρώτο σημείο ότι δεν είναι αξιόπιστα τα δεδομένα για το θέμα της πειρατείας ε, στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας διότι προέρχονται κυρίως από έρευνες που γίνονται από τις επιχειρήσεις και συνεπώς οι εκτιμήσει αρνητικού αντικτύπου που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί η πειρατεία ή η παραποίηση στον τομέα δεν είναι αξιόπιστες. Θα πρέπει στην γνωμοδότησή μας να είναι σαφές ότι μας ενδιαφέρει να προσδιοριστεί αυτό. Να υπενθυμίσω ότι το 2012 δημιουργήθηκε ένα παρατηρητήριο το οποίο συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πιο αξιόπιστα δεδομένα. Έχει κάνει έρευνα και μετά ε, από τι έρευνε προκύπτει ένα δεύτερο σημείο, το παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ευαισθησία των νέων σε σχέση με τη χρήση περιεχομένου πολιτισμικού με μη σωστό και παράνομο τρόπο ε, χέρι χαμηλής ευαισθησίας γιατί είχαμε και την ιστορία της δωρεάν πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να καθορίσουμε πιο καθαρά τη σχέση μεταξύ των επενδύσεων στη δημιουργικότητα ε, για την ίση αμοιβή των ε, δημιουργών αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την ευαισθητοποίηση των νέων, ώστε να υπάρξει μέλλον στους κλάδους αυτούς και να διευρύνουμε τους τρόπους πρόσβασης με νέες προσφορές, με διάφορα business model, ώστε ο κλάδος αυτός να είναι πιο ανοιχτός προς τους χρήστες. Γι' αυτό το παρατηρητήριο και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο της Επιτροπής προτείνουν να ξεκινήσει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με ε, πρόσθετες δράσεις με τέτοιο σκοπό. Άλλο θέμα θα θυμάστε ότι είχαμε μια σημαντική οδηγία για τα ορφανά έργα τέχνης και για την πιθανή πρόσβαση σε αυτά τα έργα κυρίως από ερευνητές, ε, φοιτητές, πανεπιστημιακούς Χρειάζεται λοιπόν περισσότερη ελευθερία σε αυτόν τον τομέα και είναι κατανοητό. Αλλά αυτό πρέπει να εξισορροπείται με την νόμιμη χρήση ε, η οποία θα πρέπει να είναι πιο ανοιχτή. Ε, η επένδυση στην έρευνα θα πρέπει επίση να παράγει και κάποια έσοδα, Αλλιώ δεν γίνεται επανεπένδυση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το θέμα ε, θα πρέπει να αντισταθμιστεί κάπω με κάποια στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξορρόπηση. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. έχετε το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις παρεμβάσεις σας. Πιστεύω ότι όλα όσα άκουσα μπορώ να τα συμπεριλάβω στο τελικό σχέδιο της γνωμοδότησής μου. Και τώρα θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα και να κάνω και κάποιες διευκρινήσεις για την πρώτη παράγραφο για τα δεδομένα. Δύο ερωτήσεις μου υπευλήθηκαν, τι εννοούμε κτλ. Ακούστε. Δεν έχουμε ούτε ακριβή ούτε αξιόπιστα δεδομένα. Αυτό όμως είναι στη φύση των πραγμάτων. Μιλάμε εδώ για αθέμητες πρακτικές. Ξορισμού λοιπόν δεν καταγράφονται. Άρα δεν μπορούμε να μετρήσουμε επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Όμως, στην περίπτωση της διανοητικής διοκτησίας, τα πράγματα διαφέρουν από τον τομέα των φαρμάκων, για παράδειγμα. και μιλώ για τον τομέα της ε, επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάποιοι κλάδοι ε, καταφεύγουν σε υπερβολές για το τι συμβαίνει στον κλάδο τους για να ασκήσουν πιέσεις και να υπάρξει αυτό το νομικό πλαίσιο. Αν αυτό το κάνει κάθε κλάδος, ε, καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα φυσικά και δεν είναι αξιόπιστα, είναι φουσκωμένα, είναι υπερβολικά. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε πάντως για να έχουμε μια αξιόπιστη βάση δεδομένων. Έχοντας πάντα κατά νου ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στην τελειότητα. Αλλά ζητώ ένα τέτοιο μηχανισμό. Αυτό εννοούσα στην παράγραφο αυτή. Είναι δύσκολο. Πώς να το πω. Σίγουρα η βιομηχανία, η κλάδη μπορούν να μας δώσουν τα πιο αξιόπιστα δεδομένα. Γιατί αυτοί ενδιαφέρονται πιο πολύ βέβαια για το τι συμβαίνει. Τώρα, έγιναν κάποιες ερωτήσεις για το άνοιγμα. Openness. δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε είτε το ένα είτε το άλλο άκρο. Δηλαδή, από τη μία όλα ανοιχτά, όλα ελεύθερα και δεν χρειαζόμαστε πνευματικά δικαιώματα και η άλλη, το άλλο άκρο όλα πρέπει να την χάνουν τις ε, αυστηρότερες να τις προστασίες. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή, τη μέση οδό. για τα πνευματικά δικαιώματα, πνευματική ιδιοκτησία. Η Επιτροπή Πολιτισμού Πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε προς την κατεύθυνση της ώστε να τρώμε μεγαλύτερης δημιουργίας. Να μπορούν και να κερδίζουν χρήματα οι καλλιτέχνες, αλλά να χρησιμοποιούν και έργα τέχνης που έχουν δημιουργηθεί παλαιότερα. Βέβαια, ε, ξεπερνά τις προσωπικές μου δυνάμεις. Ε, δεν μπορώ να βρω την τέλεια διατύπωση μέσα στις λίγες γραμμές που μπορώ να συντάξω για το θέμα αυτό. Τώρα η επιβολή δικαιωμάτων ματικής ιδιοκτησίας και κίνδυνη, η αντιμετώπιση κινδύνων. Το καλύτερο παράδειγμα για μένα δεν είναι ο τομέας ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά ο τομέας των φαρμάκων. Απομιμήσεις, παραποιημένα φάρμακα μπορεί να είναι επικίνδυνα να είναι επιβλαβή για την υγεία. Άλλο αυτό και άλλο η χρήση ενός εμπορικού σήματος. Παράνομη χρήση. Ο κλάδος έχει την τάση να ασχολείται με αυτά τα θέματα για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό. Απλά Υπάρχει και η πτυχή του καταναλωτή που πρέπει να τον προστατεύουμε από την κατάχρηση, αλλά αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ είπα να μην με αυτά τα δύο. Ευχαριστούμε κύριε Ρέιμον. Σίγουρα θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε τροποποιήσεις, τροπολογίες, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 12 το μεσημέρι στις 22 Ιανουαρίου. Επειδή εδώ λέει ότι ο κύριος Ζαν Μπερζεβά βρίσκεται εδώ από την Κομισιόν, θέλετε να πείτε δυο λόγια γι' αυτό. Ε, μπορείτε να πάρετε το λόγο αν επιθυμείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ικανοποίησή μου που η Επιτροπή αυτή θα συμβάλλει με μια γνωμοδότηση στο έργο της Επιτροπής, ε, της ουσίας Επιστροπής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά τα δεδομένα να βρει κανείς ε, αντικειμενικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο φτιάξαμε το παρατηρητήριο το οποίο καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες. Εμείς ε, ενθαρρύνουμε διαρκώς τον κλάδο να παράσχει τα δεδομένα με αντικειμενική μορφή αλλά ακούγοντα διάφορες απόψεις εδώ στην Επιτροπή εξακολουθεί να είναι πρόβλημα η αξιολόγηση μιας παράνομης δραστηριότητας αλλά εμείς σίγουρα καλωσορίζουμε περισσότερη αντικειμενικότητα στα δεδομένα αυτά και εκεί επικεντρώνεται το έργο του παρατηρητηρίου. Κάτι άλλο το οποίο αναδεικνύεται από όλα αυτά είναι ότι σε αυτό το σχέδιο δράσης θα χρησιμεύσει να, δώσουμε, να υπογραμμίσουμε το ζήτημα της ε, δεύτερη επιμέλειας. Δόθηκε το παράδειγμα του όταν χρησιμοποιούνται καλλιτέχνες τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας κατά των καλλιτεχνών, κατά της ε, θεμητής αμοιβή ε, στον τομέα των έργων ε, υπάρχει και το θέμα της δέωσης επιμέλειας για τους διάφορους διαμεσολαβητές. Όχι μόνο στις πλατφόρμες που υπάρχουν online, αφορά όλους τους διαμεσολαβητές στην αλυσίδα αξιών. Η παροχή υπηρεσιών πληρωμής, για παράδειγμα, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν κάτι περισσότερο για να παρεμποδίσουν τις πληρωμές ε, προς site παρανομών δραστηριοτήτων. Χαιρόμαστε λοιπόν που η Επιτροπή αυτή θα συμβάλλει στην έκθεση του Κοινοβουλίου. Αυτά ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας περάσουμε τώρα στην επόμενη έκθεση της οποίας η συγγετρία είμαι εγώ. Εν συντομία πρόκειται για την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Ρέτζη για την πρόθεση της οικονομικής και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση. Ξέρετε ότι τον περασμένο Ιούλιο η Κομισιόν δημοσίευσε την έκθεση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής έκθεση που πρέπει να εκπονείται κάθε τρία χρόνια και αφορά τις πρόοδους που έχουν επιτευχθεί. Η έκτη έκθεση της Κομισιόν αναλύει την κατάσταση σε αυτές τις εποχές κρίσης, τι έχει γίνει με το θέμα της συνοχής σε αυτές τις εποχές κρίσης και αναφέρει πως είναι σημαντικό να συνεχιστούν αυτές οι παραβάσεις ακόμα και με τις τροποποιήσεις που έχουμε ζητήσει εμείς ως Κοινοβούλιο και ζητά τονίζει πόσο σημαντικό είναι αυτό για το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και ε, παρουσιάζει και τις δυσκολίες ε, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πρόθεση αυτής της πολιτικής. Κατά την απόψή μου, στη γνωμοδότησή μου, συγγνώμη, προσπάθησα να συμπεριλάβω κάποιες λίγες γραμμές σε κάποιες λίγες γραμμές ε, του στρατηγικούς στόχους της Ευρώπης 2020 στόχους όπου πρέπει να συγκλίνουν τα διευθυντικά ταμεία και η συνοχή. Για να αντιμετωπιστεί η ενέργεια των νέων, μέσω για παράδειγμα της ε, μείωση της αποχώρησης, της πρώτης αποχώρησης από το σχολείο, η συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ε, η διαβίου εκπαίδευση των ενηλίκων. Επίσης, εξυγχρονισμός των συστημάτων παιδείας και ενίσχυση μέσω εδαφικών συνεργασιών, της συνεργασίας μεταξύ έρευνας, παιδείας και απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα. Το άλλο θέμα είναι το ζήτημα των διαρθρωτικών ταμείων που προβλέπεται και στην εγγύηση για τους νέους. Και ε, ο συντονισμός με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και οι εταιρικές σχέσεις που μπορούν να δημιουργηθούν ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως ε, αυτή η εγγύηση και των διορθωτικών ταμείων ώστε να δημιουργηθούν υποδομές που θα βοηθήσουν ε, όλες τις πτυχές αυτού του θέματος. Κάτι άλλο, το να αναγνωρίσουμε την ε, πλήρη συμβολή και τις δυνατότητες του πολιτισμού για την οικονομική ανάπτυξη όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, τουριστικών τον πολιτιστικό τουρισμό και τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας. Όπως βλέπουμε ε, σε όλα αυτά τα σημεία υπόαση τόσο μικρών επιχειρήσεων, νέων μικρών συστατών επιχειρήσεων. Όλα αυτά για τη βελτίωση τη ποιότητα και των θέσεων εργασία. Το άλλο σημείο είναι το θέμα τη αστική διάσταση πέραν τη περιφερειακή αυτής της οικονομικής ανάπτυξης μέσω του πολιτιστικού τουρισμού. Και φυσικά τα μέσα Αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων των ευρωπαϊκών πόλεων. Αυτά συνοπτικά. Αν θέλετε να σχολιάσετε, να προσθέσετε κάτι, όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα παρά τους περιορισμούς ε, χώρου του κειμένου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει, τι μας επισημαίνουν οι διάφορες χώρες τα ανώτατα όρια που επιβάλλονται ε, για τον πολιτιστικό τουρισμό στα διάφορα διαρθρωτικά ταμεία. Γι' αυτό θα ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες ε, και από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο σε όποιον το επιθυμεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. για την ανάπτυξη του θέματος. Σημαντικό θέμα. Μιλούμε για 8 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία προορίζονται για τον πολιτισμό. και με κίνητρα για τη δημιουργία απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού. Για κάθε 15 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι δημιουργηθούν 1.000 θέσεις απασχόλησης. Εδώ πρέπει βέβαια να μας απασχολήσουν δύο θέματα. Αφενός βλέπουμε τις προσπάθειες για αποτελεσματικότερη διαμόρφωση των δαπανών αυτών, αποδοτικότερη δηλαδή. Από την άλλη μεριά έχουμε τις νομοθετικές διαδικασίες, κανονισμούς που εν τέλει καθιστούν δύσκολο να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα συνοχής στην Ευρώπη. Δηλαδή, ως παράδειγμα, η θέσπιση πολλού υψηλού συντελεστού ΦΠΑ για τις οικοδομές, για εμβληματικά κτίρια και τα οποία έχουν υπαχθεί στους καταλόγους της UNESCO. Ε, ως αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής καθιστάμεθα μάρτυρες μιας αύξησης κατά 10% των δαπανών του κόστους της ανακαίνησης των κτίριων αυτών. Άλλο παράδειγμα. Μπαίνουν περιορισμοί στις δαπάνες των ταμείων όχι μόνο για την πολιτιστική κληρονομιά αλλά και για την βελτίωση τουριστικών υποδομών και καλλιτεχνικών σχολών. Μίλησα για μια οροφή 5 εκατομμυρίων ευρώ για την ε, δισεκατομμύριο μάλλον για την πενταετία 2015-2020. Τώρα το συνολικό ποσό θα είναι των 7,3 δισεκατομμυρίων. Χάνονται λίγο εδώ οι διαστάσεις. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει την ευρύτερη εικόνα, να επανεξετάσει την προσέγγιση που έχει επιλέξει και να εξασφαλίσει ότι θα έχουν απόδοση τα χρήματα αυτά που θα δαπανηθούν, που θα επενδυθούν, γιατί αλλιώς θα χάσουμε την ευκαιρία να επιφέρουμε βελτιώσεις στον τομέα του πολιτισμού. Και αυτό αφορά και τα έργα που υποστηρίζει η UNESCO ή τέλο πάντων που έχει περιλάβει στου καταλληλού η UNESCO και όπου έχει μπει οροφή 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι παράλογο. Τέλο, η πολιτιστική συνοχή στην Ευρώπη ξαναμπαίνει εδώ ως θέμα. Και έρχομαι στο θέμα των καλλιτεχνικών σχολών ή σχολών τέχνης. Κάτι το οποίο βελτιώνει την καλλιτεχνική παιδεία του κόσμου, των πολιτών. ώστε να έχουν μεγαλύτερη επαφή με το πολιτιστικό γίγνεσθε ανά τον κόσμο. Αυτό είναι σημαντικό. Όταν λοιπόν θα συζητήσουμε την έκθεση θα φροντίσω να καταθέσω και τροπολογίες. Ευχαριστούμε για τα όσα επισημάνατε. Μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι ευχαρίστως θα προσθέσω αυτό το σημείο και με δική μου τροπολογία. Ε, um, Ευχαριστώ πολύ. Το σχέδιο γνωμοδότησης της ε, συγγητριάς μας φαίνεται να αποτελεί μια περιεκτική γνωμοδότηση για τη στρατηγική για το 2020. Έχει κάποιους βασικούς στόχους να μειωθούν κατά 10% ποσοστά της σχολικής εγκατάλειψης πρόωρα και ένα άλλο ποσοστό 40%. Νομίζω ότι η δεύτερη παράγραφος είναι πάρα πολύ σημαντική διότι για να μην έχουμε αναντιστοιχίες μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας θα πρέπει να επενδύσουμε στον εξυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων. Πρέπει επίσης να επιδείσουμε στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνα ε, και απασχόλησης σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και επίσης να προωθήσουμε τη διασυνεργική συνεργασία. Συμφωνώ πλήρως με την ιδέα να συμπεριληφθεί το πρόγραμμα εγγύηση για την νεολαία. Είναι σημαντικό κομμάτι του όλου πακέτου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την υλοποίηση της εγγύησης για την νεολαία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι καλό λοιπόν και αυτό το σημείο για τις τελευταίες δύο παραγράφους που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά και τους τομείς ε, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Σημαντικές παράγραφοι. Ως Επιτροπή πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει το πλήρε δυναμικό του πολιτισμού που συνεισφέρει και στην οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση τη κοινωνική συνοχή. Η Κομισιόν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία τη πολιτική συνοχή για να βελτιώσει και να αυξήσει τι θέσει εργασία στον τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών για να μπορέσουν αυτές να ανθίσουν στον ψηφιακό κόσμο. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε μια νέα όθηση στην πολιτική συνοχής, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της νέας περίοδου προγραμματισμού, πρέπει να βελτιστοποιήσουμε λοιπόν το δυναμικό αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η κυρία Μωράν Σάρτια, που με μεγάλη χαρά ξαναβρίσκουμε στην Επιτροπή Πολιτισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τη βάση των προτάσεών σας και ειδικότερα με την παράγραφο 1 όπου υπενθυμίζετε τους στόχους του Ευρώπη 2020 όσον αφορά τον πολιτισμό, την παιδεία, την κατάρτιση και την ενημέρωση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ωστόσο, σε δύο σημεία Υπάρχουν δύο σημεία που πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να προσθεθούν σε αυτή την παράγραφο. Λέτε ότι 15% των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχουν σε δραστηριότητες παιδείας και κατάρτισης διαβίου. Αυτό όμω θεωρώ εγώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να εξελίσσονται αυτές οι δραστηριότητες παιδείας και κατάρτισης, διαβίου κατάρτισης, ε, να βασίζονται σε δύο παιδεία σημαντικά όχι να γίνεται πλέον θεωρητική παιδεία, αλλά πρακτική. Γι' αυτό πιστεύω είναι σημαντικό να προσθέσουμε τον όρο επικύρωση των δεξιοτήτων ε, για την επαγγελματική κινητικότητα. Το δεύτερο που μου φαίνεται σημαντικό είναι ότι πρέπει να επισημάνουμε την επικύρωση της αποκτηθής σας εμπειρίας αυτή η αποκτηθήσα εμπειρία επιτρέπει στους απασχολούμενους να έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα εντός των επιχειρήσεών τους ή μεταξύ επιχειρήσεων. Η καταπολέμηση λοιπόν της ανεργίας θα βασιστεί σε αυτούς τους δύο μοχλούς την επικύρωση των δεξιοτήτων και την επικύρωση της αποκτήθησα εμπορίας διότι εκεί μαγειρεύεται η κοινωνική συνοχή και μου φαίνεται πολύ σημαντικό και πιστεύω θα φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα η σύγκληση αυτών των δύο σημείων. Το δεύτερο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι η παράγραφος 3. Αναφέρεται την εγγύηση για την νεολαία που όπως ξέρουμε αποτελεί το μοχλό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων. Δυστυχώς η εγγύηση αυτή για τους νέους συνοδεύεται από ένα δεύτερο μοχλό την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Και ξέρετε κυρία Πρόεδρε πόσο μεγάλη σύγχυση έχει δημιουργηθεί μεταξύ αυτών των δύο της εγγύησης για τους νέους και ε, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Δεν μπορούμε λοιπόν να βάζουμε πρωτοβουλία εγγύησης για τους νέους γιατί θα διατηρήσουμε αυτή τη σύγχυση μεταξύ της εγγύησης για τους ε, νέους και ε, πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε ότι χαιρετίζουμε την εγγύηση ε, το, για τους νέους, για την καταπολέμηση της ανεργίας, ενισχυμένη στις πιο φτωχές περιοχές από την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων ενισχύει την εγγύηση για τους νέους στις περι... Ε, περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία των νέων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προσέχουμε τι λέξεις χρησιμοποιούμε γιατί σε όλα τα επίπεδα παρατηρώ ότι υπάρχει τεράστια σύγχυση. Πρέπει λοιπόν η Επιτροπή μας που εμπλέκεται τόσο πολύ σε αυτό το θέμα να είναι απολύτω σαφή. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πρόεδρε εκ των προτέρων για τα όσα θα κάνετε για να ξεκαθαρίσετε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ. Τα λαμβάνω υπόψη. Η κυρία Λιμπάτσκα. Mm, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την γνωμοδότηση αυτή και για το γεγονός ότι επισημαίνεται ότι η βάση για την μεταφική και κοινωνική συνοχή μεταξύ άλλων περνά και από την δυνατότητα έβρεσης εργασίας. Όσο πιο χαμηλά είναι τα ποσοστά ανεργίας, τόσες, ε, τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες ε, για, και οι πιθανότητες για μεγαλύτερη συνοχή. Πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε την ανεργία και ένας ε, καλός τρόπος είναι να εισαγάγουμε αλλαγές στο σύστημα. Και μιλώ για το εκπαιδευτικό σύστημα, που είναι υπεύθυνο αρμόδιο για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Αλλά εμπειρία αποκτά κανείς μόνο όταν δουλεύει. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα πρόσβασης στην κατάρτιση. Και αυτό εξαρτάται και από την ε, ικανότητα των επιχειρήσεων να υποδεχθούν σε προγράμματα μαθητείας, για παράδειγμα, ή κατάρτισης επιχειρησιακής τους νέους. Θα έχουμε έτσι και μεγαλύτερη κινητικότητα και ανταλλαγές που θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από την πολιτική συνοχή ή από το πρόγραμμα Εράσμους. Ή ίσως και από την εγγύηση για την νεολαία. Για όλα αυτά θεωρώ ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για την Πολωνία ξέρω ότι κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ θετικό. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ σημαντική σας πρόταση. Περνάμε στην Πέτρα, Κάμερεβερτ και μετά έχουμε άλλους διαμελητές. Ευχαριστώ, θα είμαι και σύντομη άλλωστε, αφού πρώτα βέβαια ευχαριστήσω για το έγγραφο. Νομίζω ότι στο λίγο πράγματι περιθώριο που σου δίνεται περιέλαβες όλα τα πιο σημαντικά που έχει να πει η Επιτροπή Πολιτισμού. Για την παράγραφο 4 έχω μια ιδέα που μπορεί ίσως να περιληφθεί και αυτή. Όλες γνωρίζουμε ότι ο πολιτισμός και η δημιουργία καλλιτεχνικών έργων συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην απασχόληση. Γνωρίζουμε επίσης ότι και με το πρόγραμμα Viewer μόνο ελάχιστη συμβολή μπορούμε να προσφέρουμε στο πολιτιστικό γίγνεσθε. Παρόλα αυτά ήμασταν πολύ ικανοποιημένες που στο παρελθόν μπορέσαμε να βάλουμε επενδύσεις στον πολιτισμό και στα διαφθορτικά ταμεία. Κοινωνικό κλπ. Και από τα χρήματα αυτά να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν και πολιτιστικά έργα θα ήταν σωστό να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως περί τα τέλη του έτους ή αρχές του επόμενου έτους, να κάνει μια προσωρινή έκθεση, σχετικά δηλαδή με το πώς εποφελούνται οι χώρες μέλη από τις νέες αυτές δυνατότητες προσφέρουν το Κοινωνικό Ταμείο, το Περιφερειακό Ταμείο για να κάνουν επενδύσεις στον πολιτισμό, στις τοπικές κοινότητες, στις περιφέρειες, αν δηλαδή πρόκειται για ένα εργαλείο, αυτό που δημιουργήσαμε, που πραγματικά χρησιμοποιείται από τις τοπικές κοινότητες, από τις περιφέρειες. Στη δική μου, στο δικό μου land, στη δική μου δηλαδή ομοσπονδιακή, στο δικό μου ομοσπονδοκρατήδιο, αυτό γίνεται. Θα ήθελα να μάθω πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε άλλες χώρες μέλη, σε άλλες περιφέρειες, αν δηλαδή εποφελούνται των κονδυλίων αυτών για να προωθήσουν επενδύσεις έστω και μικρέ στο χώρο του πολιτισμού. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα είπατε. Θα σα απαντήσω σίγουρα Έλγα Τρούπελ και μετά ο κ. Σιβέτη. Έλγα Τρούπελ. Να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εμείς παραπονούμαστε ότι οι creative industries δεν έχουν ενταχθεί επαρκώς όσο θα έπρεπε στην Ευρώπη 2020. Το ίδιο ισχύει όμως και την πολιτική συνοχής. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο πολιτιστικός κλάδος πρέπει να χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Συνοχής. Υπάρχουν πρόσθετες δυνατότητες εκεί και πρέπει να εφαρμοστεί. Δεύτερη ιδέα, με την διδημοποίηση πόλεων του In Cities, έχουμε συλλέξει πολλές θετικές εμπειρίες. Τώρα όμως έχει κάπως μειωθεί ο προϋπολογισμός για αυτά. Επειδή όμως αυτό έχει σχέση με την ενδυνάμωση του κόσμου, το empowering people δηλαδή, και με την εξασφάλιση μιας κοινωνικής συνοχής, ίσως υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουμε ώστε η δημοποίηση πόλεων να προωθηθεί περισσότερο. Να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι δηλαδή να αναπτύξουν κοινά έργα. Και διαρωτώ με αν αυτό είναι δυνατόν μέσα από αυτή την πολιτική συνοχή να χρηματοδοτηθούν περισσότερες δραστηριότητες Twin Cities. Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα σχόλιά σας. Πριν απαντήσω θα ήθελα... Α, συγγνώμη, ο κύριος Λιούερ. Δεν πειράζει, λέει ο κύριος Λιούερ. Ευχαριστώ. Είναι κουραστική και μεγάλη η σημερινή ημέρα, κυρία Πρόεδρε. Να σχολιάσω τα σχόλια που έγιναν από τον κύριο Τζαμπάσκη, το σκιώδη συγκεκριτή της ομάδας μας. Σας ευχαριστούμε για την εκθέσή σα και λέει ο ίδιο ότι η ενεργεια των νέων είναι μια από τι μεγαλύτερε προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη σήμερα. Συνεπώ πρέπει να ληφθούν μέτρα επένδυση σε παιδεία που να σχετίζεται με τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Να προσθέσω και εγώ ω συντονιστή ECR ε, για την Επιτροπή Ρέτζη, όπω και αυτήν εδώ, να πω λοιπόν ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι μίλησαν για την αποτελεσματικότητα των δαπανών και πολύ σωστά. Διότι η προσέγγιση του έχουμε ένα πρόβλημα και βάζουμε σε αυτό ένα σωρό λεφτά των φορολογουμένων ε, για να φέρει αποτέλεσμα, δεν φέρνει τελικά αποτέλεσμα. Μερικές φορές ε, αν αυτά τα χρήματα δεν είχαν έρθει στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είχαν δαπανηθεί καλύτερα. Αν ε, όπως είχε πει ο Γλάθ, είχαν παραμείνει στις τσέπες των ανθρώπων εντός της ελεύθερης αγοράς τα είχαν δαπανηθεί καλύτερα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να τα δούμε κάπως αλλιώς τα πράγματα εδώ ως Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, ειδικότερα από εκπαιδευτική άποψη για την υποστήριξη της πολιτικής συνοχής. Οι χώρες τους που μπήκαν από το 2004 και το 2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταλαβαίνω ότι χρειάζονται τη χρηματοδότηση του Ταμείου συνοχή, Επειδή οι περισσότερε από αυτέ χρειάστηκε να αποτινάξουν το ζυγό του καταπιεστικού κομμουνισμού που γνωρίζουν πολλά μέλη της Επιτροπής εδώ, πολλά από τα οποία δεν είναι παρόντα. Ορισμένες όμως χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1981 και ακόμα λαμβάνουν τεράστια κονδύλια χωρίς να εφαρμοστεί και πολύ συνοχή μετά από 34 χρόνια. 34 χρόνια είναι μια ολόκληρη καριέρα, μια ολόκληρη σταδιοδρομία. Χρειαζόμαστε λοιπόν πλήρη ανασχεδιασμό της ε, ε, συνοχής και η παιδεία, η εκπαίδευση θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού. Αναμένω λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να δούμε πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Ζητώ ακόμη συγγνώμη. Και πάλι συγγνώμη κύριε Λιούερ ε, κύριε Κάλμαν από την... Ε, η κυρία Κάλμαν από την ε, Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, καλωσορίζουμε την γνωμοδότηση. Εκπροσωπώ την ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ εκπαίδευση και πολιτισμό. Συμφωνούμε με τα περισσότερα επιχειρήματα που ακούστηκαν και εγώ θα ήθελα να τονίσω τη σημασία του δυναμικού της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο των διαθετικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, από την πλευρά των επενδύσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και από την πλευρά του πολιτισμού. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η πολιτική συνοχή ήδη έχει συνεισφέρει τα μάλα και στο προηγούμενο ε, πλαίσιο προγραμματισμού 2007-2013. Η εκτονιστέρων αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη και σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα. Για το μέλλον, δηλαδή για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, παρακολουθείτε τις διαπραγματεύσεις από ό,τι ξέρω οι μεταρρυθμίσεις ε, έχουν ένα πολύ σημαντικό άξονα, δηλαδή την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική και του στόχους Ευρώπη 2020 και στήριξη και των βασικών ε, στόχων ε, που αφορούν άμεσα κάποια από αυτούς την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό για επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Έχουμε και διαπραγματεύσεις ε, για τις μελλοντικέ ε, συμφωνίες σύνδεσης, έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις αυτές και ήδη βλέπουμε κάποια αποτελέσματα. Ξέρετε ότι μετά την έγκριση του νομικού πακέτου ακολουθεί μια ακόμη φάση που είναι η διαπραγμάτευση των ε, μελλοντικών συμφωνιών εταιρική σχέση, συγγνώμη, όχι σύνδεση, εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτηθούν. Ξέρουμε ήδη ότι εκπαίδευση και κατάρτιση έχουν 32,8 ε, ε, δισεκατομμύρια προπολογισμό, επενδύσεις, για επενδύσεις μιλάω, είναι τεράστιο το ποσό. Είναι το μεγαλύτερο σαν χρηματοδοτικό εργαλείο για την ε, επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τα 26 δις προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και τα 6,3 θα επενδυθούν σε εκπαιδευτικές υποδομές. Αυτά τα γνωρίζουμε ήδη για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υποδιαιρέσεις ε, από κάτω, δεν μπορώ να σας δώσω πιο αναλυτικά στοιχεία, γιατί οι διαπραγματεύσεις για τα επιχειρησιακά προγράμματα δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, άρα θα γνωρίζουμε περισσότερα σε μεταγενέστερο στάδιο. Γι' αυτό και δεν μπορώ να σας δώσω και νούμερα για τον πολιτιστικό και δημιουργικό κλάδο μόνο σε επίπεδο επιχειρησιακών προγραμμάτων θα μπορούμε να έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα. Αλλά για τον όγκο βλέπετε ήδη ότι είναι μεγάλος όγκος, μεγάλος ο και από τη δική μας πλευρά, γάμα δέλτα εκπαίδευση πολιτισμός, βοηθούμε τη γάμα δέλτα Ρέγγιο και τη γάμα δέλτα απασχόληση στην ε, εκτίμηση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων για να έχουμε και μια διασύνδεση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και τα διαθροτικά ταμεία αλλά και τις προτεραιότητες ή τη 2020 και τα κονδύλια του προπολογισμού που αφορούν ε, την, ε, τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Θα ήθελα να δώσω έμφαση και σε μια άλλη διάσταση του θέματος. Επενδύσει ε, στην εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω των εθνοτικών ταμείων. Αυτό δεν είναι βασικό για τους βασικούς μόνο στόχους, αλλά και για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Χαιρετίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι αναφέρετε το θέμα αυτό στην γνωμοδότησή σας. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω και το ρόλο των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ως παραγόντων πρόληψης της ανεργίας των νέων. Θέλουμε να έχουμε βιώσιμα αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, άρα πρέπει να εξυγχρονιστούν ε, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για να μην αναπαραγάγουμε ε, ανεργία μεταξύ των νέων. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να υπενθυμίσω τις προθεσμίες για τις τροπολογίες. 27 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι και να απαντήσω σε κάποια από τα σημαντικά σας σχόλια και τις προτάσεις σας και τις προσθήκες που προτείνετε που εγώ είμαι διατεθειμένη να δεχθώ ορισμένα από αυτά τα σχόλια θα αποτελέσουν το αντικείμενο τροπολογιών εφόσον τα συμμεριζόμαστε στον κύριο Ντοριευσκή ήθελα να πω ότι ακριβώς μιλάμε για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα το έχουμε ξανασυζητήσει μπορούμε να το εμβαθύνουμε και στην Επιτροπή Πολιτισμού όταν θα συζητάμε τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης ε, που θα ε, ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες. Στο πλαίσιο τώρα των καθημερινών γραμμών ε, που υπάρχουν για τα διαρθρωτικά ταμεία δεν αναφέρεται ακριβώς το όριο των 5 εκατομμυρίων, απλά γίνεται αναφορά σε ένα γεγονός που κατά την κρίση μου πρέπει να συζητηθεί λέει in any case, σε κάθε περίπτωση, οι πολιτιστικέ υποδομές μεγάλη κλίμακας σίγουρα δεν είναι προτεραιότητα και πρέπει να εξαιρεθούν από τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Περιφερειακή ανάπτυξη. Κάτι που πρέπει να εμβαθύνουμε και να συμπεριλάβουμε στην έκθεσή μας ω στοιχείο προς διευκρίνηση σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Ρέτζη. Όσον αφορά την ενίσχυση του πολιτισμού ως βασικής διάστασης για την επίτευξη της συνοχής, της απασχόλησης και της καταπολέμησης της ενεργείας των νέων, συμφωνώ απόλυτα. Θα το ενισχύσω στο κείμενο στην κυρία, Σαρτιέ, στην κυρία Μόνα Σαρτιέ να πω ότι αν εσείς, ε, ε, βασικά εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει περιορισμός λέξεων ε, στην έκθεση αυτή. Ο σκοπός είναι να πούμε ότι η εγγύηση για την νεολαία ενισχύει σίγουρα τη δέσμευση κονδυλίων για τους νέους που υπάρχουν στα διαρθρωτικά ταμεία. Μπορούμε να το πούμε ακόμη πιο καθαρά και να υπενθυμίσουμε, γιατί μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο το κοινωνικό ταμείο, να υπενθυμίσουμε όχι τόσο τον ορισμό των συστημάτων παιδείας, αλλά την ενίσχυση των δεξιοτήτων για την εργασία και την επαλήθευση αυτών των δεξιοτήτων. Στην κυρία Λιμπάτσκα θα ήθελα να πω ότι η πρόταση σας είναι πολύ καλή. Να θυμίσω ότι το σύστημα EURES που δημιουργήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να ευνοήσει την έρευνα και τις σχετικές προγράμματα μαθητείας και εργασίας Οπότε θα λάβουμε την πρότασή σας, τη δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Κέντρου Ενημέρωσης για τις ασκήσεις και τις μαθητείες. Στην Πέτρα Καμερεβέρτ θέλω να πω ότι για τα όσα είπατε, ε, εγώ συμφωνώ μαζί σας. γιατί να μην έχουμε οριζόντια συνεργασία με τις άλλες επιτροπές. Πιστεύω και με την Επιτροπή Ρέτζι θα πρέπει να αναπτύξουμε σχέσεις. Είναι απολύτως εφικτό, αρκεί να το αποφασίσουμε, να κάνουμε μια πρώτη συνεννόηση με την Επιτροπή Ρέτζι για να επαληθεύσουμε τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων στον τομέα του πολιτισμού. Έλγα Τρίπελ, συμφωνώ, η αδελφοποίηση των πόλεων κάτι που έχει οριμάσει όπως και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες ε, έχει οδηγήσει σε νέες προσεγγίσεις της αστικής ε, ε, κουλτούρας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε, να εκπονήσουμε κάποια σημαντική πρόταση, να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το δίκτυο EuroCities που περιλαμβάνει και της EuroCities πολιτισμού. Η επόμενη συνάντηση θα λάβει χώρα στο Τωρίνο στο πλαίσιο αυτό, καλό θα ήταν να αναπτύξουμε και την πρόταση που κάνατε εσείς προηγουμένως. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν φυσικά για τις διευκρινήσεις. Θα θέλαμε, καθώς θα προχωρούν ε, οι συνεργασίες, να μας ενημερώνετε για το τι κάνετε εσείς και για το που βρισκόμαστε όσον αφορά τόσο τους πόρους για την παιδεία όσο και τους πόρους για τον πολιτισμό στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Εγώ βλέπω πολύ θετικά τα σχόλιά σας. Ξέχασα μια επίκριση του κυρίου Λιούερ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι τα διαρθρωτικά ταμεία δεν έχουν δαπανηθεί πάντα σωστά, όχι μόνο σε μια χώρα, αλλά σε πολλές. Ωστόσο, πιστεύω ότι με τους νέους κανονισμούς θα έχουμε μεγαλύτερο προσανατολισμό προς την δημιουργία κινήτρων και αντικινήτρων κυκλοφορώντα τι καλύτερε πρακτικέ και τι καλύτερε εμπειρίε σε αυτόν τον τομέα, μπορεί να χρησιμεύσει ώστε να αρθούν οι δυσκολίε σχεδιασμού που υπάρχουν, απλοποιώντα τα ταμεία. Κάπως έχουν βελτιωθεί τα πράγματα σήμερα για πρώτη φορά στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Έχουμε μια 5, ένα ποσοστό 5% απευθείας ε, αφιερωμένο στις αστικές περιοχές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για, την για τον τοπικό προγραμματισμό και σχεδιασμό. Καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι απόλυτα τους κινδύνους που αναφέρετε, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική επενδυτική για μεγαλύτερη ανάπτυξη και απασχόληση. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε τον συνάδελφο Μισελ Διακόνου που θα παρουσιάσει τη γνωμοδότηση για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Είχαμε και μια καταπληκτική ακρόαση από αυτού του θέματος. Εγώ δεν βρισκόμουν εδώ, αλλά την παρακολουθούσα μέσω διαδικτύου. Εγώ ακούω τα πάντα. Ήταν εξαιρετική ακρόση και σας συγχαίρω όλους σας και όλους μας για την εξαιρετική ανάλυση. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Nu știu de ce am senzația că, de fapt, de două zile, aceste două zile, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις δύο ημέρες φαίνεται ότι συζητάμε μόνο ουσιαστικά για την πολιτιστική κληρονομιά. Έτσι, δεν είναι το μόνο αυτό. Όμως, όταν ένα έργο τέχνης ε, φτάνει σε ένα επίπεδο ποιότητας και ηλικία συγκεκριμένη, τότε κατατάσσεται πλέον ε, στην πολιτιστική κληρονομιά. Σας ευχαριστώ που με εμπιστευτήκατε για να συντάξω αυτή την έκθεση. Αυτό που θέλησα να κάνω ήταν να συμπεριλάβω όσο το δυνατόν περισσότερες απόψεις και από την Ιταλική Προεδρία, την Επιτροπή Περιφερειών που γνωμοδότησε, το Συμβούλιο και βέβαια έλαβε υπόψη και την άποψη της κοινή γνώμης των εμπειρογνωμόνων και θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω μάλλον τους συντονιστές που δέχθηκαν για να, τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και θέλω να ευχαριστήσω και τη γραμματεία που ανέλαβε τη διεξαγωγή αυτής της, την οργάνωση αυτής της ακρόασης. Περιμένω όλοι να συνεισφέρουν στη βελτίωση της έκθεσης, σκιώδεις εγκητές και μη. Όλοι θέλω να συνεισφέρουν. Και καλό θα ήταν να γίνει μια συνεδρίαση όλων των σκιωδών εισηγητών, αν συμφωνείτε βέβαια, μπορώ να έρθω εγώ σε επαφή με τη γραμματεία και να το κανονίσω. Να πω τώρα τι θεωρώ σημαντικό. Καταρχάς, χρηματοδότηση της πολιτικής κληρονομιάς μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Είναι το πλέον δύσκολο ζήτημα, διότι πρέπει να το αντιμετωπίσει κανείς με την μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. η κρίση που πλήττει εδώ και περισσότερο από έξι χρόνια την Ευρώπη έχει πλήξει και τα ταμεία, τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για την πρόσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι εθνικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να προστατεύσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. Υπήρχαν πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούσαν τη διαφύλαξη πολιτική κληρονομιά και δεν υπάρχουν πλέον δυστυχώ. Έχουμε τώρα τη Δημιουργική Ευρώπη, την Ευρώπη 2020 με κονδύλια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουμε και κονδύλια από την Αλία και την Γεωργία. Δυστυχώ όμως βλέπουμε να λιγοστεύουν όλο και περισσότερο αυτά τα κονδύλια. Πάντως εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας και οι τοπικές και περιφερειακέ περιφερειακές αρχές δεν τα γνωρίζουν αυτά τα εργαλεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια πάρα πολύ καλή ιδέα να τα συγκεντρώσει τα εργαλεία αυτά σε έναν κατάλογο, σε ένα έγγραφο. Σε αυτό το έγγραφο εξηγεί ποια είναι όλα αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία, όμως δυστυχώς είναι μόνο στα αγγλικά αυτό το έγγραφο. Και είναι και άκρος τεχνικό. Χρησιμοποιεί τη γλώσσα που χρησιμοποιούν ε, τα θεσμικά όργανα. Δεν είναι απλό. Δεν είναι κατανοητό. Θα ζητούσα λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιεί λιγότερο τεχνική γλώσσα, ε, να είναι πιο εύληπτο αυτό το εγγραφό που είναι τόσο καλό και αν είναι δυνατόν και σε άλλες γλώσσες για να μπορεί να διαδοθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Τα μέτρα λιτότητα σίγουρα είχαν καταστρεπτικές, ε, καταστροφικές συνέπειες και φαίνεται και το λέω και στην έκθεσή μου. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών υπήρξαν πολύ καλές ε, πρακτικές στον τομέα του πολιτισμού και ανταλλαγή αυτών. Δεν υπάρχει όμως ε, μια μελέτη ευρωπαϊκή η οποία να βασίζεται σε αυτά τα δεδομένα. Επειδή λοιπόν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα, θα παρακαλέσω τους εκπροσώπους της να δουν. Υπάρχει βάση δεδομένων γι' αυτό και αν όχι να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα Τρίτο θέμα. Συμμετοχική διακυβέρνηση. Δεν χρησιμοποιείται και τόσο συχνά αυτός ο ώρας τελευταία. Στόχο πάντως έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην επικοινωνία. Είναι ένα μοντέλο και δημοκρατικό, αλλά βελτιώνει και την οικονομική κατάσταση. και στην εποχή αυτή των ισχνών αγελάδων σίγουρα μπορεί να βοηθήσει τον πολιτιστικό κλάδο να ορθοποδήσει. Καλό είναι λοιπόν να έχουμε ε, και ανταλλαγή απόψεων για το πώς μπορούμε καλύτερα να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Ένα πολύ γνωστό, επιτυχημένο παράδειγμα είναι αυτό των Ιταλών ηθοποιών που ανέλαβαν την διαχείριση ενός τοπικού θεάτρου και με τον τρόπο αυτό το έσωσαν το θέατρο αυτό που θα έκλεινε αλλιώς. ηθοποιοί γενικά είναι ευαίσθητοι σε τέτοιες ε, ενέργειες και δράσεις, διότι βλέπουν ε, ότι η τοπική κοινωνία με τις ε, δράσεις της μπορεί να αντιμετωπίσει τις απειλές και κάποια συλλογικά μέτρα που λαμβάνονται. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξτάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας νομικών μέσων που θα νομιμοποιούν τέτοιου είδους πρακτικές που μέχρι τώρα παραμένουν άτυπες. πρέπει οι πολίτες ε, να οικειοποιηθούν την πολιτιστική κληρονομιά. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς. Ε, είναι μια γερμανική πρόταση. Βέβαια πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις. Ε, αυτό το ευρωπαϊκό έτος θα πρέπει να έχει τον κατάλληλο προϋπολογισμό και κατά δεύτερον τα κράτη-μέλη πρέπει να συμμετέχουν από την αρχή, δηλαδή να υποβάλουν σχέδια, προγράμματα για να εμπλουτίσουν και να κάνουν ε, πραγματικότητα τελικά αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Είναι μια ιδέα που οριμάζει σιγά σιγά και νομίζω ότι μπορούμε να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Ένα άλλο ζήτημα που ήθελα να αναφέρω εδώ είναι η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Πολυάριθμες ευκαιρίες μας προσφέρει η η νέα τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία και μπορούμε να τι εφαρμόσουμε στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι τεχνολογικές και μη καινοτομίε. και η κινητοποίηση των νέων, η παρακίνηση των νέων να συμμετάσχουν είναι όλα προς όφελός μας. Υπάρχει μεγάλη τεχνολογική καινοτομία στις χώρες μέλη. Θα έπρεπε να την εκμεταλλευτούμε. Έχουμε την τεχνολογική πλατφόρμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της οποίας ε, θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί η ψηφιοποίηση. Δεν ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια όμως. Γνωρίζουμε ότι ιδέες υπάρχουν, αλλά πρέπει να βαθύνουμε περισσότερο. Επόμενο σημείο να πούμε ότι η κληρονομιά η πολιτιστική έχει βέβαια πρώτα απ' όλα πολιτιστική αξία. Αλλά και οικονομική. Είμαστε σε εποχή κρίσης και μιλάμε μόνο για οικονομία, άρα να μην πούμε και όλα εδώ ότι πέραν της καλλιτεχνικής αξίας πολιτισμός είναι κλειδί για την όθηση της οικονομίας και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ιδίως σε παραδοσιακά επαγγέλματα που αλλιώς χάνονται. Και για να χρησιμοποιήσω και ένα οικονομικό επιχείρημα, μπορώ να πω ότι το βασικό πρόβλημα στις μέρες μας είναι η απόλυτα εργασίας στον πολιτιστικό κλάδο. Που αν στηριχθεί, ο πολιτιστικός κλάδος δηλαδή, μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα της απόλυτα εργασία. Ολοκληρώνοντας, θέλω να αναφέρω ένα θέμα που μπορεί να μην φαίνεται επίκαιρο, εγώ όμως νομίζω ότι είναι μονίμως επίκαιρο. Και μιλώ για τη διακίνηση έργων τέχνης, που είναι απειλή για τον πολιτισμό και έχει πολύ μεγάλη σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις που έχουμε με άλλες χώρες. Αυτά προς το παρόν. Με ανυπομονησία περιμένω τα δικά σας σχόλια. Ευχαριστούμε ειλικρινά. Αυτή είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Σας παρόν να είστε σύντομοι διότι στη συνέχεια έχουμε τη σημαντική έκθεση για τη ε, Δημιουργική Ευρώπη. Ό,τι έχετε να πείτε, πείτε τα γρήγορα. Μόργανο, παρακαλώ. Ε, βλέπω πολύ κόσμο θέλει να μιλήσει. Έχουμε λίγο χρόνο, λοιπόν. Παρακαλώ, Μόργανο. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή που παρέθεσε πολλά σημεία προς προβληματισμό, τα οποία συμμερίζομαι. Αναμένουμε να διαβάσουμε το σχέδιο έκθεσης για να εκφράσουμε την πολιτική μας εκτίμηση. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδιαίτερα τη διαφύλιξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς υπό την ευρεία έννοια. Δεν είναι ε, μία από τις οδούς για την επανεκκίνηση της οικονομίας της Ένωσης, αλλά η κύρια οδός. Οπότε επιτρέψτε μου μια παρένθεση που πιστεύω δεν είναι άσχετη. Δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τα τραγικά γεγονότα στο Παρίσι που μας απέδειξαν δυστυχώς όχι μόνο πως η κοινωνία και η δημοκρατία μας είναι ευάλωτες αλλά κυρίως ότι υπάρχει κάτι περισσότερο το οποίο πρέπει να κάνουμε. Ότι κάτι δεν λειτουργήσε το σύστημα που χρησιμοποιούμε για να εκτιμήσουν πολλοί νέοι την πολιτιστική μας κληρονομιά, οδηγώντας ε, σε κοινωνικά προβλήματα και περιθωριοποίηση. Αυτό το λέω για να πω ότι παρά τις δεσμεύσεις των κρατών για την παιδεία, είδαμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να εξετάσουμε μόνο αυτή την πτυχή για να συμφωνήσουμε όλοι ότι η είναι απαραίτητο να βρούμε νέους τρόπους μετάδοσης ε, και διαφήμισης ε, της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο για τη διαφύλαξή της αλλά και για την πρόθεση της δημοκρατικής μας κοινωνίας ε, για την καταπολέμηση κάθε μορφής μυσαλλοδοξίας και για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου σε γενικότερο επίπεδο. Είναι κατεπήγον πέραν του εκπαιδευτικού συστήματος να προωθήσουμε τη γνώση των υπολογιστών και τη σωστή χρήση των πόρων που προέρχονται από κάθε περιοχή της Ευρώπης. Να προωθήσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα εφαρμοστούν όσο καλύτερες είναι οι πρακτικές έρευνας και στα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όπως υπογραμμίστηκε και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πολιτιστική μας κληρονομιά, ο εξαιρετικός χαρακτήρας ε, της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ε, ηλικής και άειλης, ε, καθεδρική ναή, αλλά και φυσικά τοπία, γλώσσες, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Είναι σίγουρα ο μεγαλύτερος μας θησαυρός κάτι πολύτιμο που εκπροσωπεί την ταυτότητα, την ιστορία μας, την αίσθησή μας ότι ανήκουμε κάπου για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι. Ένα κεφάλαιο λοιπόν το οποίο αναφέρεται εδώ στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στο κείμενο του εισηγητή μας οδηγεί σε ένα καθήκον, καθήκον να τα προστατεύσουμε όλα αυτά και να τα αναδείξουμε. Σήμερα βλέποντας αυτό το γεγονός που μας δυσκόλεψε τόσο πολύ. Πρέπει να συνδέσουμε την οικονομία με τον πολιτισμό και να ενώσουμε τις πτυχές της τεχνολογίας, του πολιτισμού, της κοινωνίας και της οικονομίας σε και σε μακροοικονομικό επίπεδο. Πρέπει να επενδύσουμε στους ανθρώπους, στην κουλτούρα με μια προσέγγιση που δεν μπορεί να είναι ίδια με την σημερινή προσέγγιση. Με τη μέχρι τώρα προσέγγιση πρέπει να δούμε πιο πέρα. Θα πρότεινα αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου και του συστήματος διακυβέρνησης και των συστημάτων διοίκησης ολόκληρου του πολιτιστικού πλούτου μια διαφορετική προσέγγιση από τους πολίτες αλλά και την συνέστηση των οικονομικών δυσκολιών που θα πρέπει να μας οδηγήσουν σε συνεργασίες μεταξύ ιδιωτικού, ε, που ε, αποδεικνύουν ότι η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ήταν ένα σφάλμα. Υπάρχουν κάποια νούμερα σήμερα που μας λένε πολλά. Να δώσω ένα παράδειγμα ως εισηγητής ε, του σχεδίου γνωμοδότησης για τις προκλήσεις του τουρισμού στην Ευρώπη υπενθυμίζω ότι η Ευρώπη είναι ένας από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίω. Ο τουρισμός είναι βασικός τομέας ε, στην οικονομία της Ευρώπης 5% του συνολικού ΑΕΠ και απασχολεί 12 εκατομμύρια ανθρώπους περίπου και περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω εδώ είναι ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιστοιχεί στο 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού. Γνωρίζοντας λοιπόν τη στρατηγική διάσταση και τις δυνατότητες του τομέα αυτού, επιβάλλεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μην προχωρήσουμε άτακτα και χωρισμένοι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε τις, συνεργα... συνέργειες. Πρέπει να υλοποιήσουμε τον ε, οριζόντιο χαρακτήρα όλων των πολιτικών της Ένωσης με μεγαλύτερες συνέργειες και συνεργασία μεταξύ διαφορών τομέων του τουρισμού, της εκπαίδευσης, του περιβάλλοντος, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής ανάπτυξης και της φορολογίας. Επιτρέψτε μου μάλιστα να σας αναδείξω, την, να, να σας παρουσιάσω την αξία, τη μακροπρόθεσμη αξία που θα έχει ε, αυτή η εστίαση στην πολιτιστική κληρονομιά, μακροχρόνια. Όπως ανέφερα στην αρχή λοιπόν, αναμένω μαζί με την ομάδα να εκτιμήσουμε τις προτάσεις του εισηγητή. Είμαι βέβαιος ότι η κοινή ευαισθησία που χαρακτηρίζει τα μέλη της Επιτροπής αυτής εδώ του Κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας, θα μπορέσει να οδηγήσει σε μια ευρέως ε, ε, ε, συμπεφωνημένη θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολύ δομημένη ήταν η παρουσίασή σα και δεν ήθελα να σα διακόψω. Σα ευχαριστούμε για τη σημαντική σα συμβολή. Στρογεύσκη, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μία πρόσκληση, δύο σχόλια, μία σύσταση. Πρώτο σημαντικό στοιχείο είναι το εξή. Ω τώρα στην Ένωση, δυστυχώ, δεν υπήρξε ποτέ σύστημα το οποίο να διατηρεί σε περιπτώσεις θεομηνιών, καταστροφών, σεισμών κλπ. τα μνημεία. Πολλά μνημεία έχουν καταστραφεί μετά από πλημμύρες, σεισμούς ή πυρκαγιές. Είναι πολύ σημαντικό στις περιπτώσεις αυτές να μπορεί να προσφέρεται πραγματική αποτελεσματική υποστήριξη. Διότι ο χρόνος αντίδρασης μετά από σεισμό ή πυρκαγιά και ούτω καθεξής έχει κέρια σημασία για να μειωθεί το κόστος και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της στήριξης. Το είδαμε το πρόβλημα αυτό στην Ασσιζή, αλλά το είδαμε και στις φωτιές στην Σλοβακία, επίσης μετά από πλημμύρες και στην Ουγγαρία το ίδιο. Τρομερές απώλειες η μνημεία. Πρώτο σχόλιο λοιπόν είναι η βοήθεια που πρέπει να προσφέρεται σε περιπτώσεις θεομηνιών. Για τη διατήρηση των μνημείων. Έχουμε βάσει δεδομένων που περιλαμβάνουν τα μνημεία στι χώρε μέλη. Αυτό που είναι σωστό, ωστόσο που έχετε δίκιο δηλαδή, είναι ότι δεν έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επίπεδο τη Ένωση για να ενσωματωθούν όλε αυτέ οι τράπεζε δεδομένων. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα καταγραφή των μνημείων έτσι ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί το σύστημα και να είναι τα δεδομένα συγκρίσιμα και δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε όλη την Ένωση. Τρίτο σχόλιο, ψηφιοποίηση. Πάλι στον χώρο των μνημείων. Οι χώρες μέλη χρησιμοποιούν διαφορετικά στάνταρτ. Διαφορετικές τυποποίησεις. Για να χρησιμοποιηθούν λοιπόν αυτά για την εκπαίδευση των νέων και των παιδιών, αυτό τελικά καθιστά αδύνατον να χρησιμοποιούν τα δεδομένα δηλαδή για την εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε λοιπόν οι ίδιες προδιαγραφές για όλες τι χώρε μέλη. Έτσι ώστε να μην χάνονται και τα κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διατήρηση των μνημείων. Τέλος, πάλι για τα μνημεία και στην Ευρώπη αλλά και εκτό αυτή. είναι πολύ χαμηλή η αποτελεσματικότητα των ε, στηρίξεων που δίνουμε. Για παράδειγμα, το Μουσείο του Κάιρο και της Αλεξάνδρειας. Στην ε, Κωνσταντινούπολη επίσης. Πολλά χρόνια δουλειά χάθηκαν. Γιατί η ποιότητα των έργων είναι πολύ χαμηλή. Των έργων υποστήριξης. Πρέπει λοιπόν να αναλύσουμε καλά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ταμεία έτσι ώστε να μην χάνονται τα κονδύλια. Σε δύο εβδομάδες θα εγκαινιάσω έκθεση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιάζω τα επιτεύγματά μας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και υποδομών. Θα είναι η μέρα Τρίτη και ώρα 18 το απόγευμα. Προσκαλείστε όλοι. Θα είμαστε εκεί δίχως άλλο ο συνάδελφος κ. Ευχαριστώ. Και εγώ κυρία Πρόεδρε δεν θα μιλήσω για τα θετικά στοιχεία της ανακοίνωσης και τα όσα ανέπτυξε ο εισηγητής γιατί βεβαίως υπάρχουν τέτοια και είναι πολλά. Χαίρομαι για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαι άλλωστε νέος Ευρωβουλευτής και θεωρώ ότι η ανακοίνωση αυτή αποδίδει μεγάλη σημασία και στον πολιτισμό και στον ρόλο που παίζει αυτό και στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική. Βεβαίω, είπαν και άλλα οι προηγούμενοι συναδελφοί μου όπω για ψηφιοποίηση, για οργάνωση μουσείων, ανταλλαγή εμπειριών με άλλε χώρε. Όλα αυτά είναι βέβαια πολύ σημαντικά. Εγώ θα ήθελα να συναγάγω ένα γενικότερο συμπέρασμα. Νομίζω ότι η Επιτροπή Πολιτισμού θα πρέπει να είναι και τόπος όπου μπορούμε να προβληματιστούμε γενικότερα πάνω στον ρόλο του πολιτισμού και για το τι σημαίνει πολιτισμός και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον πολιτισμό. Νομίζω τα έγγραφά μας πρέπει να περιλαμβάνουν μια προσέγγιση στον πολιτισμό. Αυτή που βλέπω τώρα ωστόσο με ενισχύει κάπως. Κάποιοι από τους προηγούμενους ομιλητές ίσως έχουν μια προσέγγιση, αλλά λίγο, λίγοι τέλος πάντων αναγνωρίζουν τη σημασία του πολιτισμού. Δεν αρκεί να προσέχουμε τα μνημεία του πολιτισμού. Ο πολιτισμός δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο διαχείρισης όπως οποιοδήποτε άλλος οικονομικός κλάδος και βεβαίως σωστό είναι αυτό. Και καλά κάνει και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο τέτοιας μεταχείρισης. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και σωστά βέβαια λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν υπάρχει αντίθεση μεταξύ, να έχω σε αντίφαση δηλαδή οι εθνικές με τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες αλλά εγώ διαρωτώ με εάν δεν είναι αλήθεια ότι το γεγονός ότι θέλουμε να οργανώσουμε, να χρηματοδοτήσουμε και να υποστηρίξουμε τον πολιτισμό, μήπως αυτά στην ουσία υπονομεύουν τα εσωτερικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού. Η ποικιλία, η πολυφωνία μπορεί να είναι και πηγή εντάσεων. Δεν μπορούν όλα να οργανωθούν, δεν μπορούν όλα να μπουν στα ίδια σχήματα. Κανένας μάνατζερ, κανένας πολιτικός δεν μπορεί να βγει να πει ποιο είναι το πραγματικά καινοτόμο στοιχείο του πολιτισμού. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε αυτά. Ποιος είναι ο ρόλος του πολιτισμού στην Ευρώπη. Αυτά δεν άπτονται απαραίτητα των όσων πράττουν ε, θρησκευτικές ομάδες ή ομαδε ομάδες μεταναστών κλπ. Στην Πολωνία συζητούμε τα θέματα αυτά πολύ. Για παράδειγμα και τη σχέση μεταξύ Πολωνών και Γερμανών για τους εκτοπισμένους από την Πολωνία μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. Αυτά όμως δεν περιλαμβάνονται στο έγγραφο γιατί το έγγραφο όλο μιλεί για εναρμόνιση, για συγκέντρωση. Ας μην αυταπατώμεθα. Η παραπάνω χρηματοδότηση, η αύξηση τη χρηματοδότησης δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εναρμόνιση. Η συμφιλίωση είναι κάτι, μια φυσική οδός πρέπει να ακολουθούμε, αλλά δεν πρέπει να οδηγήσει στην εξόντωση της δημιουργικότητας. Ας το έχουμε αυτό υπόψη μας όλες και όλοι. Και ας συγκρατήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλες αυτές τις προσπάθειες που καταβάλει για συγκέντρωση και διαχείριση των πάντων από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι θα πρέπει μάλλον να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις, τις αντιθέσεις ως πηγή δημιουργικότητας. Ο πολιτισμός δεν είναι πάντα κάτι που ε, μπορεί να το παρουσιάσει κανείς έτσι ωραιοποιημένο στα μουσεία. Είναι καμιά φορά και ο αγώνας, ε, είναι εξέγερση. Ε, κοιτάξτε τον Χάιντεγκερ. Καμιά φορά προβάλλουν ιδέες που ίσως μας φαίνονται και απαράδεκτες, αλλά μπορεί να είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικέ. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στο έγγραφό μας. Και αυτά βέβαια έχουν και επιπτώσεις στον τρόπο που διαχειριστούμε τον πολιτισμό. Αφού όλοι δεχόμαστε εδώ την ελεύθερη οικονομία της αγοράς, πρέπει να δεχτούμε και την ελευθερία του πολιτισμού. Ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφοι, τι ενδιαφέρονται αυτά που είπατε. Μαραγάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το πώς εστιάζει την εκθεσή του ο συνάδελφος. Είναι πολύ καλή προοπτική και η δόμηση της έκθεσης που είναι σημαντικό και νομίζω ότι είναι πιο γενικό το θέμα. Ναι, μεν μπορεί να φαίνεται ότι εστιάζουμε σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, την προστασία δηλαδή της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά είναι πιο γενικό το ζήτημα. Το ακούσαμε και από τον προλαλήσαντα. Τι θα πει η Ευρώπη, πώς μπορούμε να δημιουργούμε και ταυτόχρονα να σεβόμαστε κτλ. Έχουμε σύμπτωση απόψεων λοιπόν, έχουμε και τα θέματα της ψηφιοποίησης, ανταλλαγής ε, πρακτικών, τοπικό επίπεδο κτλ. Θα έχουμε δυνατότητα να σχολιάσουμε, να προσθέσω όμως και ορισμένα ζητήματα ή κάτι ε, που προηγείται αν θέλετε. Τι θα κάνουμε εδώ, θα συζητήσουμε το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε με κάποιες αποχρώσεις ε, και με κάποια συγκεκριμένα σημεία. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν το status quo να προσαρμόσουμε αυτή την πολιτική που ήδη υπάρχει ή αυτό που θα κάνουμε τελικά είναι ότι θα δούμε ότι υπάρχει ένα σημείο, ε, μια καμψή αν θέλετε, και θα πρέπει να περκεράσουμε αυτή την καμψή και να στραφούμε προς το μέλλον και να μην περιορίσουμε στο παρόν. Έχω και κάποια ερωτήματα. Αν όλοι συμφωνήσουμε ότι και τα οικονομικά μεγέθη και η οικονομική δραστηριότητα και η σημασία επίση που έχει ο πολιτισμό και ο τουρισμό για την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργία θέσεων κλπ. Αν συμφωνήσουμε ότι έχουν όλα αυτά σημασία, ταυτότητα ε, και συμφιλές με το παρελθόν κτλ. Ναι, καλό αυτό, αλλά λείπει και η μελλοντική προοπτική. Να δώσουμε έναν ορίζοντα ε, μελλοντικό και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα συστήματα τη πολιτιστική κληρονομιά. Και υπάρχει και μια κατάφορη αντίφαση. Εάν εμεί ε, διακηρύσουμε την σημασία την οικονομική αυτού του φαινομένου, Πώ δεχόμαστε τόσο παθητικά αυτή την όλο και λιγότερη απόδοση πόρων και κονδυλίων σε αυτό το τόσο σημαντικό κατά τα άλλα τομέα και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο όλο και μειώνονται οι δαπάνες για τα πολιτισμικά. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Μια ερώτηση τώρα που με απασχολεί και νομίζω ότι και όλους πρέπει να μας απασχολήσει. Γιατί να μην μιλάμε υπό όρους ευρωπαϊκών πολιτιστικών αγαθών. Έχουμε τοπικά, εθνικά και παγκόσμια πολιτιστικά αγαθά, όχι ευρωπαϊκά όμως και δεν υπάρχει και ευρωπαϊκή προστασία αυτών των πολιτιστικών αγαθών. Πολλά πολιτιστικά αγαθά παγκόσμιο ενδιαφέροντος μεταξύ αυτών, όπως της UNESCO για παράδειγμα, ε, έχουμε τέτοια μνημεία που ούτε τα προστατεύουμε και πολλές φορές τα εγκαταλείπουμε. Στη χώρα μου έχω τέτοια παραδείγματα. Άρα ευρωπαϊκό πολιτιστικό αγαθό. Είναι μια έννοια που θα έπρεπε να διερευνήσουμε. Θα πρέπει επίση να δούμε αν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και περιφερειών. Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν αρμοδιότητε. Γιατί να περιμένουμε, γιατί να φιλτράρουμε, να δούμε το αποτέλεσμα ε, μετά από τη αμεσολάβηση παρέμβαση των κρατών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει άμεση σχέση περιφερειών με Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη έννοια που νομίζω ότι πρέπει να την ε, αναπτύξουμε. Υπάρχει στην έκθεση, αλλά να αναπτύξουμε περαιτέρω. Ιστορικές διαδρομές διεθνείς, διασυνοριακές. Όχι μόνο στο ιστορικό μιας χώρας με τοπικό, ιστορικό ενδιαφέρον, από πλάι και τα λοιπά, αλλά που θα μπορέσουν να προσδιορίσουν την ευρωπαϊκή ιστορία. Μια άλλη έννοια που αυτή δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση. Πρέπει όμως να συμπεριληφθεί. Ευρωπαϊκή πόλη ε, που έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά Ιταλία. Η Ιταλία είναι ένας κατάλογος μακροσκελέστατος με τέτοιες πόλεις και από την πλευρά της ποιότητας ζωής και της αρχιτεκτονικής, της διάρτημης κτλ. Της, σύμφωνα, της ρημοτομίας. Νομίζω ότι πρέπει να συμπεριλάβουμε στην πολιτική κληρονομιά αυτές τις πόλεις. Έκτον, ο πολιτισμός ζει από τις παροχές, από τους πόρους, από τα ταμείο συνοχής ε, κτλ. Όχι όμως από ένα άμεσο και μετρήσιμο κονδύλι. Αποκλειστικά δηλαδή αφαιρωμένο για τα θέματα του πολιτισμού, που θα έπρεπε να υπάρχει όμως. Τέλος, και σχετίζεται αυτό με τα προηγούμενα που είπα, Νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε μια σαφή στρατηγική με ευρωπαϊκούς στόχους και μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα μας δώσουν τη δυνατότητα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο να αξιολογήσουμε, να μετρήσουμε το τι συμβαίνει, ποιοι ήταν οι στόχοι μας, ε, ποιους πετύχαμε, όπως κάνουμε τα προγράμματα περιφερειακής σύγκλησης για τις περιφέρειες κτλ. Και να είναι και αποτελεσματική κατανομή αρμοδιοτήτων σε εθνικό, τοπικό επίπεδο, επίπεδο πόνο κτλ πολλά υποσχόμενο το μέλλον. Ε, νομίζω ότι μπορούμε με την έκθεση αυτή να προσφέρουμε προς τη θέμενη ευρωπαϊκή αξία, όπως λέμε. Ευχαριστώ. Thank you. And... Ευχαριστούμε. Ε, Τζούλη. Word, παρακαλώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, κάνοντας ένα σχόλιο. Να αναφερθώ στο, για, ποιο λόγο, στο για ποιο λόγο πρέπει να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό πρέπει να γίνει με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των διαφορών λαών της Ευρώπης που ενδεχομένως να έχουν διενέξεις μεταξύ τους. ώστε το μέλλον να είναι πιο ασφαλές, πιο ειρηνικό. η πολιτιστική κληρονομιά έχει ένα παίξει σημαντικό ρόλο. Θα μας βοηθήσει να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο για όλους. Από, από αυτού λοιπόν θα ήθελα να προτείνω πρέπει να επενδυθούν χρήματα σε υπευθύνους εκπαίδευσης στο να διατηρούνται, το να διατηρούνται οι συλλογές και να διατηρούνται για πρόσβαση στο κοινό δεν βοηθά πρέπει να έχουμε κάποιους που να ερμηνεύουν αυτές τις συλλογές ώστε είναι να καταλαβαίνουν το παρελθόν και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για το δίκτυο οργανώσεων Ευρωπαϊκών Μουσείων στην Πολόνια τον Νοέμβριο. Πριν από αυτό έκανα κάποια έρευνα στη δική μου περιοχή για να δω τα δικά μας μουσεία, τα μικρά και μεγάλα, τα χρηματοδοτούμενα από τις τοπικές αρχές ε, ή άλλους χρηματοδοτούμενα, να δω λοιπόν τι κάνουν για να συνεργαστούν μαζί με τις κοινότητες ώστε να γίνουν πιο κατανοητές οι συλλογές τους και ε, υπάρχουν πολλές βέλτιστες πρακτικές εκεί. Ο καλύτερος τρόπος για να εξοικονομήσουμε χρήματα είναι να μοιραστούμε ιδέες, γνώσεις, ε, πρακτικές και να επενδύονται τα χρήματα στους σωστούς τομείς. Να φροντίσουμε λοιπόν να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους για να αξιοποιούν αυτές τις συλλογέ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό θα ήθελα να ε, ε, λάβει περισσότερη εστίαση. Το λόγο, ευχαριστούμε, το λόγο έχει η κυρία Σουίντροβα. Vážené kolegyně a kolegové, když eh, tuto tak Ευχαριστώ πολύ. Ε, διάβασα την έκθεση αυτή και συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι να ασχοληθούμε αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή τελικά μας φαίνει στο πυρήνα. Τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να αποκαλέσουμε πολιστικό πλούτο της Ευρώπης. Ε, Θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία τα οποία διάβασα ότι περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση και τα θεωρώ θετικά. Για παράδειγμα το γεγονός ότι η έκθεση λέει ότι θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε αναλόγως την πολιτική κληρονομιά. Δεν υπάρχει κατάλογος ευρετήριο όλων των πολιτικών έργων. Έγινε μια προσπάθεια το 2013 και έχουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα. Υπάρχουν δημόσιες ε, πηγές, δημόσιοι πόροι. Θα πρέπει όμως να ποσοτικοποιήσουμε την αξία της πολιτικής κληρονομιάς ε, και τη συνεισφορά που έχει και στην οικονομία. Αυτό πρέπει να τονιστεί στην έκθεση και είναι πολύ σημαντικό για τη μελλοντική μας δουλειά. Η έκθεση σε μεγάλο βαθμό ασχολείται με το τι κάνουμε ε, στον τομέα των επιστημών. Πώς μπορούμε τα μνημεία, τα πολιτιστικά και τις νέες επιστημονικές μεθόδους να τις χρησιμοποιήσουμε για την διάδοση του πολιτισμού. Έχουμε ε, πολύ καλές εμπειρίες. Πρέπει να διαφυλάξουμε πάντως αυτά τα μνημεία. Εκεί που βλέπω κάποια έλλειψη είναι ότι δεν δίνεται επαρκής έμφαση στα άειλα πολιτιστικά αγαθά. Κάνει λόγο βέβαια ο εισηγητής και για τα άλλα και για τα υλικά πολιτιστικά αγαθά, ε, πολιτιστική κληρονομιά λοιπόν, άειλη και υλική αλλά δεν έχουμε 100% ισορροπία μεταξύ των δύο. Δίνεται μεγαλύτερη σημασία στα υλικά αγαθά. Εγώ νομίζω όμως ότι υπάρχουν και πολλά άλλα πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν στην πολιτική και εδώ δεν αναφέρονται. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή θα έπρεπε να προσανατολιστεί περισσότερο και στην χρήση κάποιων προγραμμάτων που έχουμε αξιολογήσει ως θετικά. Ε, ε, Έχουμε ξεκινήσει και ένα πρόγραμμα για ε, την Ευρωπαϊκή Πολιστική Πατέψα από τις 17 Ιανουαρίου. Τρέχει για ένα χρόνο αυτό το πρόγραμμα. Στο Πίλσεν θα ξεκινήσει λοιπόν ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων το οποίο έχει να κάνει με την πολιτική κληρονομιά. Κάνει και συγκεκριμένε προτάσεις η έκθεση, το πώς μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ε, να αναφέρουμε και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Κάποιοι συνάδελφοι το ανέφεραν το θέμα αυτό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Η εκπαίδευση οι καλές τέχνες πρέπει να ενταχθούν σε αυτήν την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ο κ. Μαραγκάλ επίσης είπε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την έννοια ευρωπαϊκό πολιτιστικό αγαθό. Αυτό ήδη γίνεται. Νομίζω το χρησιμοποιούμε ήδη ως τίτλο, ως χαρακτηρισμό αυτό, το ευρωπαϊκό πολιτιστικό αγαθό. přístupu a tak dále. Čili rozumím tomu jeho návrhu, ale rozumím také tomu, že, že tento termín Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε όμως όταν μπορεί να προσφέρει προσθέμενη αξία. Ο Πολωνός συνάδελφος είχε μια καλή ιδέα να μας μεταφέρει. Να σκεφτούμε δηλαδή και πιο θεωρητικά τι είναι αυτό που αποτελεί πολιτισμό και τι σχέση θα έπρεπε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε να έχουμε συγκέντρωση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το οποίο προσφέρει είναι κίνητρα, προγράμματα, όπου τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να πάρουν κάποια μέτρα για να προωθήσουν τη δική τους πολιτική κληρονομιά. Δεν τους υπαγορεύεται κάτι από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Προσφορά. Μια προσφορά γίνεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο και κάποια κράτη μπορούν να αξιοποιήσουν την πολιτική κληρονομιά pro zachování a Αυτή η μέθοδος συντονισμού λοιπόν ε, νομίζω ότι πολλά μπορεί να προσφέρει για τη διατήρηση της πολιτικής Βέβαια, η πρόταση για μια θεωρητική εισαγωγή που φαίνεται σου πίσω σωστή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί όλες και όλοι είμαστε λίγο κουρασμένοι. Νομίζω ότι και άλλοι συμμερίζονται την άποψή μου όταν λέγω ότι είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Εκπροσωπούμε πολλές χώρες με ποικιλία πολιτισμών και αυτή η ποικιλία πολιτισμών είναι και από, μόνο, μόνη της ένας ελκυστικός παράγοντας. Ο κύριος Διακόνου είναι άνθρωπος της πράξης. Είναι ηθοποιός ο ίδιος. Άρα προέρχεται από το επάγγελμα και γνωρίζει την υπόθεση αυτή. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το γνωρίζει καλά. Η ψηφιοποίηση μου φαίνεται σημαντική και λογική αποτελεί και ένα τρόπο προστασίας αυτής της ποικιλομορφία των πολιτιστικών παραδόσεων και συμβάλλει σε μια καλύτερη κατανόηση του κοινού μας παρελθόντος, καθώς επίσης και μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τους γειτονές μας. Αφού μας επιτρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα τις ε, ε, παραδόσεις των γειτόνων μας, όπως είπε ο κ. Ντρογεύσκη, όταν ε, συμβαίνουν καταστροφές, θεομηνίες κλπ. Καταστρέφονται μνημεία και αυτά δύσκολα επανέρχονται. Κύριος Μαλτέζε, παρακαλώ. Δεν θέλω και εγώ να καταχρηστώ τις υπομονή των συναδέλφων. Θα περιοριστώ σε ένα σημείο από τα πολλά που θα ήθελα να αναφέρω. Θα εστιαστώ στη συμμετοχή. Χαίρομαι που ο κύριος Διακόνου ανέφερε την εμπειρία του Βαλ, όπου συμμετείχα και εγώ. Τι συνέβη εκεί. Πρόκειται για ένα ιστορικό θέατρο της Ρώμης, πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό υπήρχε ο κίνδυνος να ιδιωτικοποιηθεί, να κλείσει και μια ομάδα καλλιτεχνών, ηθοποιών, αλλά όχι μόνο αυτή, ουσιαστικά όλος ο πληθυσμός, όλοι οι κάτοικοι της γειτονιάς εξεγέρθησαν όταν άκουσαν αυτή τη λύση. Με τρόπο όμως δυστυχώς παράνομο. Δηλαδή αυτή η κατάληψη ήταν επιτυχής αλλά υπήρχε διαρκώς η απειλή παρέμβασης ε, για την εκένωση του κτηρίου πολλές τέτοιε περιπτώσεις έχουμε σε ιστορικά κέντρα στην πόλη μου, στη Ρώμη. Υπάρχει ένα ένας ιστορικός κινηματογράφος, πολύ σημαντικός, στο Τραστέβερε, στη γειτονιά του Τραστέβερε, που επρόκειτο να μετατραπεί σε αίθουσα για μπίνγκο. Και οι κάτοικοι της γειτονιάς ε, επαναστάτησαν, αντέδρασαν στην ιδέα του να αλλάξει ε, ρόλο το κτίριο ενός τόσο σημαντικού ε, κινηματογράφου για να πηγαίνουν ε, συνταξιούχοι να παίζουν bridge υπό το βλέμμα των μαφιόζων για τους ανθρώπους αυτούς. Ε, μάλιστα νομίζω ο, και η πρόεδρος της Επιτροπής, νομίζω ζει εκεί κοντά. Ε. ε να, ε, ναι, μιλήστε για τραστέβερ, ε, μένω ναι, λέει η πρόεδρος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε, να μελετήσουμε τα διάφορα μέσα για να διευκρινίσουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι κοινή. Έχουμε τεράστια πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη και στην Ιταλία. Όχι μόνο γιατί είχαμε μεγάλους καλλιτέχνες ή μεγάλους ε, χρηματοδότες αυτών των καλλιτεχνών, αλλά γιατί οι πληθυσμοί μας έζησαν, συμμετείχαν, προστάτευσαν κατά τη διάρκεια των πολέμων, των καταστροφών που έπλεξαν αυτή την Ήπειρο τα πολιτιστικά αγαθά σαν ε, ήταν ιδιοκτήτες τους. Αυτή η συμμετοχή των καταστροφων που επλεξαν αυτη την ηπειρο τα πολιτιστικα αγαθα σαν ηταν ιδιοκτητε τους αυτη η συμμετοχη λοιπον θα πρέπει να αναγνωριστεί είναι παράδοξο στη δική μου χώρα ας πούμε να σήμερα οι κάτοικοι να μην ε, λένε τη γνώμη τους για το τι θα συμβεί με ένα ιστορικό κτίριο, με ένα κινηματογράφο, με ένα ιστορικό θέατρο, κάτι που ήταν ε, σαφές κατά την αναγέννηση στη χώρα μου. Δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο του ιδεώδους της Ευρώπης όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Ευχαριστούμε, κυρία Τρούπελ. Εγώ <clears throat> ήθελα μόνο να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, παρόλο που δεν είναι κατάλληλο ένα σύντομο σχόλιο, στον κύριο Κατουμπέρσκι. Ο πολιτισμός δεν είναι πάντοτε μόνο συμπαθητικά πράγματα. Είναι και γύρω από συγκρούσεις και μπορεί να είναι και αγώνας. Από την άλλη μεριά, αυτό που αποτελεί ευρωπαϊκό επιτευγμα είναι ότι κατέστησε τον πολιτισμό καθαρά αποτέλεσμα ελεύθερης συζήτησης, ελευθερίας τύπου, ελευθερίας σκέψης. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπορέσαμε να βρούμε μια κοινή βάση συμβίωσης, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όλοι καταπολεμούμε τους εξτρεμισμούς και τον ρατσισμό. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα θεμέλιο της δημοκρατικής ζωής αλλά και του πολιτισμού. Και νομίζω ότι υπάρχουν κοινοί αγώνες και είναι καθαρό ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε ποια είναι η δημοκρατική αντίληψη για τον πολιτισμό. Και αυτό πιστεύω ότι εμείς προωθούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τα έξω είναι ότι αυτές οι αντιλήψεις, αυτή η αντίληψη, το κόνσεπτ αυτό της προβολής διάφορων οπτικών μέσα σε ένα πραγματικό γνήσιο διάλογο και ότι θα πρέπει ε, να απαγορεύεται να προχωρήσουμε προς ε, εξτρεμισμούς ή ε, και βία. Ευχαριστούμε για αυτή την τελευταία παρέμβαση της κυρίας Τρόπελ που συμμεριζόμαι πλήρως. Ήταν εξαιρετική αυτή η συζήτηση κύριε Διακόνου, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για αυτή την έκθεση που θα παρουσιαστεί 24 Μαρτίου και η ψηφοφορία προβλέπεται για τον Ιούνιο. Να δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Σερμίνα Σακητάνο από την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού αν θέλει να πει κάτι, κάποιες παρατηρήσεις ε, για την έκθεση αυτή και μετά, ζητώ συγγνώμη, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους όσοι βρίσκονται εδώ, όσους άδειξαν μέχρι τώρα, αμέσως μετά Έχουμε τον Δόκτωρ Μανέ από την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού που θα μας παρουσιάσει κάτι πολύ σημαντικό. Πώς δηλαδή προχώρα η εφαρμογή του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Ένα από τα δύο σημαντικότερα προγράμματα που έχουμε εγκρινεί εμεί. Θα σας παρακαλήσω λοιπόν να παραμείνετε στην αίθουσα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή την πρώτη παρουσίαση της έκθεσης για την πολιτική κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημειώσαμε τις απόψεις του κυρίου Διακονού και της ε, Επιτροπής Πολιτισμού σε σχέση με την ανακοίνωση της Επιτροπής. Η πρώτη απαντήση που μπορώ να σας δω. έχω πολλές απαντήσεις να δώσω, η πρώτη αφορά το ερώτημα του κυρίου Διακόνου που αφορά τον τρόπο με τον οποίο κοινοποιείται η υποστήριξη για τα προγράμματα σας και τις πολιτικές. Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Οι πληροφορίες αυτές συνοψίζονται σε δύο συμπληρωματικά έγγραφα. Το πρώτο είναι η ίδια η ανακοίνωση προς μια ενοποιημένη προσέγγιση της πολιτικής κληρονομιάς για την Ευρώπη, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει τις ευκαιρίες που υπάρχουν στι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και τα προγράμματα για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό είναι ένα πολιτικό έγγραφο, αλλά έχει συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευρέω προσπελάσιμο και κατανοητό. Προορίζεται και για το ευρύτερο κοινό και έχει μεταφραστεί σε όλε τι επίσημε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέχεια έχουμε την έκθεση χαρτογράφηση που αναφέρατε με αναλυτικές πληροφορίες για πολιτικές, νομοθεσία, προγράμματα και χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Η έκθεση χαρτογράφησης κυκλοφορεί μόνο στα αγγλικά, αλλά απευθύνεται σε ένα πιο περιορισμένο κοινό. Αποσκοπιστώ να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους και τους υπευθύνους, τους ηθήνοντες σε κάθε κράτος μέλος για τα διάφορα προγράμματα και πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο λεπτομερώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να επικαιροποιεί διαρκώς αυτή τη χαρτογράφηση. Ωστόσο, δεν ε, υπάρχει πρόθεση να μεταφραστεί σε άλλε γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πρακτικού και δημοσιονομικού λόγου, διότι είναι αδύνατο να, να μεταφράζεται έγκαιρα. Γιατί κάθε φορά που θα γίνεται μετάφραση, μετά αμέσω θα πρέπει να επικυρωποιείται, διότι τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα σε αυτόν τον τομέα. Η δεύτερη ερώτηση του εισηγητή αφορά το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ύπαρξη μιας πλατφόρμας ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα τη πολιτιστικής κληρονομιά. Με μεγάλη χαρά ενημερώνουμε την Επιτροπή σας ότι υπάρχει μια νέα πλατφόρμα διάδοσης που μόλις έχει δημιουργήσει, δημιουργήσει η Κομισιόν, βρίσκεται σε φάση υλοποίηση. Αυτή η πλατφόρμα, η Valor, εμφανίζεται ως βάση δεδομένων προγραμμάτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη και καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση ερευνών μέσω λέξεων κλειδιά. Επίση, το Συμβούλιο τον περασμένο Νοέμβριο υθέτησε ένα νέο πρόγραμμα για τον πολιτισμό, όπω γνωρίζετε, που περιλαμβάνει την πολιτιστική κληρονομιά ω μία από τι τέσσερι προτεραιότητε από το 2015 μέχρι το 2018. Το σχέδιο εργασιών προτείνει διάφορα πράγματα για τις πολι πολιτικές, ε, πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρώτη ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί με τη συμμετοχική διακυβέρνηση για την πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή νέα μοντέλα διαχείρισης ε, της πολιτιστικής κληρονομιάς. Νομίζω ότι αναφέρθηκε αυτό σε ερωτήσεις. Το Η δεύτερη συνάντηση θα αφορά την εκπαίδευση και τη μεταφορά γνώσεων για την πολιτιστική κληρονομιά. Θέλει μια πολύτιμη πλατφόρμα για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Ε, εθνικών ηθινόντων για την πολιτική κληρονομιά. Ξέρετε, στο πλαίσιο της ανοιχτής μεθόδου συντονισμού ε, θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες στην τομέα της παιδείας. Επίσης, με μεγάλη μας χαρά σας ενημερώνουμε ότι στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη έχουμε μόλις ξεκινήσει ένα πιλωτικό έργο που προωθεί την εκμάθηση μεταξύ ομοτήμων, μεταξύ περιφερειών ε, και κρατών για ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ διαφόρων τομέων ε, συμπεριλαμβάνεται και η πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο θα υποστηρίξει την ανταλλαγή εμπειριών με άμεσες επαφές μεταξύ πόλεων, περιφερειών, διοικήσεων μέσω επισκέψεων μελετών με follow-up και ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να μεγιστοποιηθούν τα ωφέλη και να υπάρχει μέγιστη δυνατή συμμετοχή σε αυτή την ευρεία διάδοση πληροφοριών. Uh, uh, Τρίτη ερώτηση για το θέμα που επισήμανε ο κ. Σίγητης στην πρόταση για την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν καλωσορίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Θα συζητηθεί εν αυτό το χρόνο. Για να ολοκληρώσω, να σας ξαναευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας οι απόψεις και τα όσα μας προβληματίσουν και τα όσα ακούσαμε εδώ θα τα λάβουμε υπόψη κατά τη διάρκεια της εργασίας μας. Αναμένουμε την έκθεση για την πολιτική κληρονομιά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος, για τις σημαντικές αυτές πληροφορίες. Μας ενδιαφέρει να μας ενημερώνετε τακτικά. Θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μας οποιαδήποτε ενημέρωση. Να σας ευχαριστήσω όλους για την ενεργό συμμετοχή σας στη συζήτηση και δίνω αμέσω το λόγο, ευχαριστώντας σας για την υπομονή σας, ε, στον Δ. Μανιέ, που τώρα θα παρέμβει για μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή για την κατάσταση πρόοδου του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη. Ευχαριστούμε και έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με την αδειά σας θα ήθελα να μιλήσω στα γαλλικά για να σας παρουσιάσω την κατάσταση προόδου της διαχείρισης του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Μετά από την πολιτική παρουσίαση που έγινε σήμερα το πρωί από τον κύριο Ναύρατζιτ, τον κύριο Επίτροπο, επιφορτισμένο με τον πολιτισμό. Η παρουσίασή μου χωρίζεται σε δύο τμήματα. Πρώτον, θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σα ε, για το πλαίσιο στο οποίο διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη και στη συνέχεια θα σα παρουσιάσω ε, κάποιες γενικές πληροφορίες για τόσα έγιναν το 2014 και για τόσα θα κάνουμε το 2015 και το 2016, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Στο πρώτο κομμάτι της παρουσίασής μου, αν μου το επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, να σας διακόψω λίγο, λέει η Πρόεδρος, φυσικά μαζί με τον κύριο Μανιέ, εκ μέρους της Γενικής Διευθυνσής Παιδείας και Πολιτισμού, θα το έλεγα μετά. σα ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί. Πρέπει να σα παρουσιάσω μαζί η κυρία Ρικάλτε από την DG Connect. Οι δύο εκπρόσωποι εδώ τη Κομισιόν ε, πιστεύουμε ότι θα μα κάνετε μια ενημέρωση πλήρη. Αυτά, αυτό θα έλεγα ακριβώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η διαχείριση του προγράμματο ε, Δημιουργική Ευρώπη χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Πολιτικό, επιχειρησιακό και διοικητικό. Το πολιτικό μας επίπεδο, πιστεύω, ε, έχει πλέον διευκρινιστεί πλήρως. Έχουμε τη νομική βάση για το πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από τον νομοθέτη στις 11 Δεκεμβρίου του 2013 και που είναι γνωστή. Έχουμε πλέον και το σχέδιο εργασία για τον πολιτισμό 2015-2018 που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο στις 25 Νοεμβρίου του 2014 και που αποτελεί την πολιτιστική στρατηγική που θα ακολουθήσουμε εμείς μέσα στην επόμενη τριετία. Και τέλος έχουμε τις, πολιτικέ τις πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές που ανακοινώθηκαν πέρυσι από τον Πρόεδρο Ζωάν Κλοντ Γιούνκερ όταν ανέλαβε καθήκοντα. Στην ε, επιστολή, αποστολή των Επιτρόπων βρίσκουμε κάποια κείμενα που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Πρόκειται για τις επιστολές του κ. Ναύρατσης που ήρθε να μιλήσει σήμερα το πρωί εδώ και του κ. Έτιγκερ του Επιτρόπου Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Να σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από αυτές τις επιστολές του κ. Ναύρατσιτ έλεγε να προωθηθεί ο πολιτισμό μέσω τη καινοτομία μεγιστοποιώντα του τομεί για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την ε, δημιουργία θέσεων εργασία, ειδικότερα ανάμεσα των, μεταξύ των νέων, για την πρόθεση τη πολιτιστική πολυμορφία και για να βοηθηθούν οι πολιτιστικοί τομεί τη Ευρώπη για να ε, αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα ακροατήρια χρησιμοποιώντα το πρόγραμμα Δημιουργική ε, Ευ... Ευρώπη για αυτό το σκοπό στην επιστολή αποστολή του κ. Έτιγκερ αναφέρεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη των δημιουργικών κλάδων και ε, ενός επιτυχούς κλάδου οπτικοακουστικών μέσων ε, με δυνατότητα πρόσβαση σε νέα ακροατήρια με τρόπο προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή και με τρόπο συνδεδεμένο με την νέα ψηφιακή αγορά. Η Κομισιόν λοιπόν που ανέλαβε καθήκοντα τον Νοέμβριο περιλαμβάνει δύο επιτρόπους οι οποίοι καλούνται να συνεργαστούν για τη διαχείριση του προγράμματος. Ο κύριο Ναύρατσιτς ε, έχει γενική συντονιστική αρμοδιότητα και ο κύριος Έτιγκερ συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την ε, ανάπτυξη των δημιουργικών κλάδων και την προώθηση της ενιαίας ψηφικής αγοράς. Ο κύριος Έτιγκερ, όπως θύμισε σήμερα το πρωί ο κύριο Ναύρατσιτς, είναι επίση αρμόδιος για το σχέδιο αναθεώρησης του πλαισίου που θα εφαρμοστεί στο copyright. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το πολιτικό πλαίσιο βάσει το οποίο παρεμβαίνουμε. Τώρα για το επιχειρησιακό πλαίσιο. Πρόσφατα άλλαξε μορφή όπως γνωρίζετε. Η Ένωση Μέσων που διευθύνει η συναδελφός μου κύριε Ρικάλντι μεταφέρθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού στη Γενική Διεύθυνση Connect. Μια τέτοια κίνηση σημαίνει το εξή, ότι υπάρχει βούληση να ευθυγραμμιστεί καλύτερα η πολιτική με το πρόγραμμα. Να γίνει μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ του υποπρογράμματος Media και του σχεδίου ενιαία ψηφιακή αγοράς. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι το πρόγραμμα έχει κοπεί στα δύο. Παραμένει ένα ενιαίο πρόγραμμα και η νομική του βάση εννοείται Εφαρμόστε εξ ολοκλήρου. Το 2014 ε, δύο μονάδες ξεχωριστές, δύο τμήματα από τη δική μας διεύθυνση διαχειρίζονταν το πρόγραμμα. Τώρα απλά τη διαχείριση έχουν δύο τμήματα που ανήκουν σε δύο γενικές διευθύνσεις διαφορετικές αλλά ε, και πάλι υπό την ευθύνη της Κομισιόν στο πλαίσιο των στόχων και προτεραιοτήτων που ορίζονται από την νομική βάση του προγράμματος. Περνάω τώρα στο διοικητικό πλαίσιο που προσαρμόστηκε σε αυτές τις αλλαγές. Αμέσως ε, προχωρήσαμε σε προσωρινές διευθετήσεις μετά την 1η Νοεμβρίου και οι δύο γενικές διευθύνσεις που είναι, αρμόδιες, που είναι συναρμόδιες πρόκειται σύντομα να συνάψουν ένα μνημόνιο συνεννόησης για να επιβεβαιωθεί η κοινή διαχείριση αυτού του προγράμματος. Και με την αδειά σας κυρία Πρόεδρε να δώσω στην κυρία Ρικάλντη το λόγο για να σας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Εγώ θα σας τα πω στα αγγλικά, αν μου επιτρέπετε. Θα σας δώσω λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο περνούμε από ένα πιο επιχειρησιακό τρόπο διαχείρισης σε ένα πιο διοικητικό. Διακόπτη η πρόεδρα. Καλύτερα παρακαλώ σβήστε το άλλο μικρόφωνο. Μάλιστα. Και υπάρχει κι άλλο ένα πίσω σας. Ωραία, ευχαριστώ. Συνεχίζω τότε να σας εξηγήσω τις διοικητικές ρυθμίσεις που έχουμε λάβει, που έχουμε θεσπίσει. Έτσι τώρα το υποπρόγραμμα το διαχειρίζεται η DigiConnect και άλλο υποπρόγραμμα άλλη ε, ε, γενική διεύθυνση χωρίς αυτό να σημαίνει ότι λειτουργούμε ξεχωριστά. Συνεργαζόμαστε στενά μέσα στα πλαίσια μιας Ομάδα ηθικών καθηκόντων, task force, που συναντάται σε τακτά διαστήματα. Να σας δώσω και λίγα παραδείγματα. Εργαζόμαστε πάνω στην σύνταξη του προγράμματος εργασιών και αργότερα βέβαια και για τις συναντήσεις των επιτροπών. Εργαζόμαστε επίσης επί των διαπραγματεύσεων με μελλοντικού συμμετέχοντες από τρίτες χώρες, επίσης για θέματα διασποράς, παρακολούθηση του προγράμματος monitoring και της συνέχειας που δίνεται, follow-up. Συνεργαζόμαστε και με τους συναδέλφους του οργανισμού για να προωθήσουμε την διαχείριση και των δύο συνιστοσών του προγράμματος και βέβαια και για τον προϋπολογισμό του 2016 καθώς και για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2015. Ιδιαίτερη προσοχή αποδώσαμε να κρατήσουμε το γραφείο σαν ενωμένη ομάδα ανθρώπων. Οργανώσαμε και πέρσι, αλλά θα οργανώσουμε και φέτος συνάντηση ώστε όσοι συμμετέχουν, όσοι μάλλον εργάζονται για τα μίδια και όσοι εργάζονται για τον πολιτισμό να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει το πρόγραμμα να συνεχιστεί ως ενιαίο σύνολο και σε λίγες εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες δηλαδή θα συνεργαστούμε πάλι μέσα στα πλαίσια της Βερλινάλες. Σας ευχαριστώ. Donc, euh, viens maintenant à la... Να έρθω τώρα στο δεύτερο τμήμα της ε, παρουσίασης. Δηλαδή, στην Επιτροπή Πολιτισμού να αναφέρουμε το τι κάναμε ε, μετά την έναρξη του προγράμματος και θα ξεκινήσω από το 2014, την πρώτη χρονιά δηλαδή. Άμεσα συναντήσαμε δυσκολίες διαχείρισης, λόγω του ότι η νομική βάση εγκρίθηκε στο τέλος του 2013. Άρα η διαχείριση του προγράμματος ξεκίνησε με μια καθυστέρηση τεσσάρων μηνών σε σχέση με τη διαχείριση την κανονική γιατί οι προκηρύξει συνήθω ε, δημοσιοποιούνται στα τέλη του χρόνου για να, τις αξιολογήσουν ο οργανισμός. Φέτος ε, ξεκινήσαμε πάρα πολύ γρήγορα τις πρώτες ε, προκηρύξεις και καταφέραμε πριν το τέλος του 2013 με κάποιους διοικητικούς, με κάποιες διοικητικές ακροβασίες τέλος πάντων που θα τις παραλείψω, δεν τις αναφέρω στην Επιτροπή σας, τα καταφέραμε. Τώρα, το 2015 για το πρόγραμμα εργασίας ήδη από, τη, από τους πρώτους μήνες ε, έπρεπε να προετοιμαστούμε για το 2015 για λόγους χρονοδιαγράμματος και έτσι δεν μπορούσαμε να υποφεληθούμε από την εμπειρία που αποκομίσαμε από το πρώτο έτος ε, για το δεύτερο έτος. Και αυτό ήταν ένας ακόμη, ένας ακόμη περιορισμός. πρώτη επιτροπή του προγράμματος ε, ε, συνεδρία το Μάρτιο του 2014 και εκεί ασχοληθήκαμε κυρίως με το πρόγραμμα εργασίας και το desk. Όπως είπε και η Λουθία, προσέγγιση των desk έγινε ικανοποιητικά. Κατά το μάλλον ή τον. Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ρυθμιστούν βέβαια. Και έχουμε λοιπόν τώρα αυτή την προσέγγιση στα περισσότερα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να τονίσω ότι την επιλογή σε όλες τις περιπτώσεις την κάναμε μέσα στο χρονοδιάγραμμα και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού. Γιατί ο κλάδο αυτό ήθελε να μπορέσει να αποφεληθεί τη χρηματοδότηση. Δηλαδή δεν είχαμε διακοπή, υπήρξε μια συνέχεια. Τήρησαμε τι προθεσμίε και χάρη στην εξαιρετική δουλειά του εκτελεστικού οργανισμού καταφέραμε να διατηρήσουμε τα πρότυπα χρηστή διαχείριση. Κάτι πολύ σημαντικό για όλα τα προγράμματα που διαχειρίζεται η Κομισιόν. Για μας η Δημιουργική Ευρώπη είναι ένα πρόγραμμα ε, στο οποίο δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κακοδιαχείρισης ή διαφθοράς. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του προγράμματος πολιτισμός και μίντια. Και θέλαμε να το διαφυλάξουμε αυτό τώρα. Το 2014 δεν χρησιμοποίησαμε πάρα πολύ τη διατομιακή πτυχή πέραν από τις δαπάνες για τα desk ή τις δαπάνες για τις δύο προεδρίες και τα έξοδα επικοινωνίας. Δεν είμαστε όμως σίγουροι τι θα γίνει με το περιπολισμό του 2015, ε, την άνοιξη του 2014. Θα θυμάστε κυρία Πρόεδρε ότι υπήρχαν προοπτικές μείωσης ε, των δεσμεύσεων ανάληψης υποχρεώσεων, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το πρόγραμμα αυτό και αυτό θέλησαμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην ρηψοκινδυνεύσουμε για τα δύο προγράμματα για να υπάρχει μια συνέχεια των επιδοτήσεων. Υπενθυμίζω ότι η καμπύλη του προγράμματος δεν είναι καθόλου ισορροπημένη, δυστυχώς. Το 2013 πολιτισμός και μίντια ήταν 186 εκατομμύρια, το 2014 179 μόνο εκατομμύρια ήταν ε, Δημιουργική Ευρώπη. Και μην πω και λίγο λιγότερο. Το 2016 θα έχουμε 196 εκατομμύρια ευρώ. Ανεβαίνουμε αισθητά. Αλλά αυτό το προφίλ δεν ευνοεί τόσο πολύ μια ευέλικτη διαχείριση των δράσεων μας. Τέλος, το 2014 δρομολογήσαμε δράσεις επικοινωνίας πάρα πολύ εντατικές, πολλές δράσεις ε, παρουσίασης σε διάφορα κρατημέλη. Ορίσαμε μια οπτική ταυτότητα για το πρόγραμμα ή στο σελίδα του προγράμματος ανανεώθηκε εντελώς και Έχουμε πλέον και μία σελίδα Facebook με 15.000 ε, ε, οπαδούς. Πρόσφατα δε δώσαμε στη δημοσιότητα ένα εργαλείο παραγωγής που λέγεται Valor και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από την ιστοσελίδα μας και εκεί να έχετε την εικόνα όλων των ε, προγραμμάτων που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Μπορεί να μην ήταν λοιπόν η τέλεια η κίνηση, αλλά θεωρούμε ότι ήταν ικανοποιητική σε γενικές γραμμές. ιδίω ό,τι αφορά ε, το, τις προκηρύξεις που ξεκίνησαν μόλις το Δεκέμβριο. Και υπήρξε μεγάλη καινοτομία και αλλαγή λόγω της αλλαγή νομική βάσης. Τηρήσαμε τις προθεσμίες, προτεραιότητά μας, πολύ σημαντική, για να μην έχουμε διακοπή της χρηματοδότησης. Και δεύτερο, η ποιότητα των έργων και σχεδίων. Εκεί δεν κάναμε κανένα συμβιβασμό. Όμως, παραμένουν κάποιες αναγκαίες βελτιώσεις. Πρέπει να είναι πιο σαφείς οι κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος, διότι για ορισμένες δράσεις οι ανάδοχοι θεώρησαν ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και πρέπει να δούμε και τι ρόλο διαδραματίζουν οι εμπειρογνώμονες στην αξιολόγηση των έργων και σχεδίων και ποιες μεθόδους εργασίας χρησιμοποιούν. Πρέπει τα desk, τα γραφεία, να δούμε ακριβώς τι ρόλο έχουν, αφού πλέον ομαδοποιήθηκαν. Πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια ε, στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών επιλογής. Πολύ σημαντικός στόχος αυτός για την πρόθεση του προγράμματος. Και τέλος, όπως υπογράμμισε σήμερα το πρωί και η κυρία Ward, σε κάποιο βαθμό θα πρέπει να επανεξισορροπήσουμε τα σχέδια συνεργασία μεταξύ μεγαλύτερη κλίμακα και μικρότερη κλίμακα σχεδίων. Και από φέτο, μάλιστα θέλουμε να τον πετύχουμε αυτό το στόχο. Τώρα, γρήγορα, γρήγορα, τι γίνεται το 2015. Σα δώσω κάποιες ε, γενικέ πληροφορίε για να συμπληρώσω τι πληροφορίε που σα έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε μια επιτροπή προγράμματο που είναι ενιαία, 28 Απριλίου συνεδριάζει και μεταξύ άλλων θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας του 2016. Θα βελτιώσουμε τις μεθόδους επιλογής με τον εκτελεστικό οργανισμό με βάση τα διαδάγματα που αντλούμε από την εμπειρία του 2014. Επίσης, θα υλοποιήσουμε καινοτόμε δράσεις στο πλαίσιο του δια... της πτυχής. Θα έχουμε το Φόρουμ του Πολιτισμού, όπως κάθε δύο χρόνια. Είναι με κοινοπραξία μεταξύ των γενικών διευθύνσεων, μια κοινή μάλλον ε, άσκηση και επίσης έχουμε προκήρυξη ε, διαγωνισμού, αλλά αυτή τη φορά με βάση το σύνηθες χρονοδιάγραμμα. Το καλοκαίρι δηλαδή και όχι στα τέλη του χρόνου θα προκηρυχθούν διαγωνισμοί. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, ξεκινάμε διαπραγματεύσεις για το εγγυητικό μέσο με τη γάμα Connect, οπότε αν δείτε την άδεια ξαναδίνω το λόγο στη συνάδελφό μου. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Όπως γνωρίζετε, η στόχη του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ε, είναι να δοθεί καλύτερη χρηματοδότηση για να μπορούν να δραστηριοποιούνται καλύτερα οι μικρομεσαίες επιχείρησεις στους τομείς αυτούς. Μέσω αυτού του μέσου στόχος είναι να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Το νέο στοιχείο του μέσου αυτού είναι η συμπριλήψη ενός συστήματος ε, δημιουργίας ικανοτήτων που είναι πολύ σημαντικό για τις τράπεζες, για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ώστε να καταλάβουν καλύτερα τα ε, εφικτά, απτά πλεονεκτήματα των σχετικών ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα. Το μέσο αυτό θα έχει προπολογισμό 121 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2016 και 2020 και αναμένουμε ότι θα έχει απόδοση 5,7 δηλαδή πιστεύουμε ότι θα αποδώσει 570 εκατομμύρια το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό ποσό οι επίσημες ε, διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει επίσημα. Ωστόσο, λαμβάνουν ήδη χώρα συζητήσεις εντατικές. Πρόθεση είναι να ξεκινήσουν επίσημα διαπραγματεύσεις κάπου το Μάρτιο και να κλείσουν, αν όλα πάνε καλά, πριν το καλοκαίρι. Έτσι θα ενεργοποιηθεί το σύστημα capacity building στο δεύτερο εξάμεινο του 2015 και η πραγματική υλοποίηση του σχεδίου θα ξεκινήσει το 2016. Και ολοκληρώνω την παρουσίαση αυτή με μια σύντομη αναφορά στο 2016 θα έχουμε το μέσω χρηματοδοτικής εγγύησης θα χρηματοδοτηθεί το τρίτο πακέτο διαγωνισμών που θα προκηρύξει κομισιόν. Φέτος νομίζω θα έχουμε και το πρώτο, ή μάλλον εκείνη τη χρονιά θα έχουμε και το πρώτο φόρουμ ε, κινηματογράφου που ανοίξει το χαρτοφυλάκιο της Γαμαλτα Connect από φέτος. Άρα θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό το πρώτο φόρμα το 2016 με βάση την ανακοίνωση που πρότεινε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέλος το 2016 ξεκινάμε την προετοιμασία της ενδιάμεσης αναθεώρησης του προγράμματος. Το άρθρο 18 που είναι η νομική βάση μας υποχρεώνει να καταθέσουμε στο ε, Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο πριν την 31η Δεκεμβρίου του 2017 αυτήν την ενδιάμεση αξιολόγηση θα απαιτήσει χρόνο, άρα θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία της αξιολόγησης αυτής ήδη από το 2016. Αυτά λοιπόν κυρία Πεδόρα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τι είχαμε να σας πούμε και βέβαια είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρουσίασή σας. Να δώσω αμέσως το λόγο σε δύο συναδέλφους που τον ζήτησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι, καταλαβαίνω φυσικά απόλυτα πρέπει να πω ότι η καθυστέρηση που αναφέρατε οφείλεται στην νέα οργάνωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω αυτό που ρώτησα και τον Επίτροπο, η ευθύνη συντονισμού του προγράμματος. Εξακολουθεί να είναι ευθύνη της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, Πολιτισμού και Παιδείας με συνεργασία της Γενικής Διεύθυνσης Connect που αναλαμβάνει το θέμα των μέσων. Υπάρχει κάποιο συντονισμό ουσιαστικά. Επίσης να ρωτήσω και κάτι άλλο σε ένα δεύτερο γύρο. Από ό,τι κατάλαβα η πρόσκληση, η, η συμφωνία που κάνετε Συγγνώμη, έχουν επιβεβαιωθεί ήδη κάποια προγράμματα το 2014. Μπορείτε να μας δώσετε και κάποιες προφορίες επί της ουσίας ε, η πρόσκληση που κάνατε, τι έγινε με τα προγράμματα, με τους πόρους. Ε? Καλό θα ήταν να μας κάνετε κάποια ενημέρωση, πιστεύω, στη δεύτερη σας απάντηση. Να δώσουμε το λόγο στους δύο συναδέλφους που θέλουν το λόγο. Yes, uh, thank you, uh, You all... Ευχαριστώ, Σίλβια. Ήδη είπατε κάποια πράγματα, αλλά εγώ θέλω να επανέλθω σε κάποιες ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον πολιτισμό. Σίγουρα λιγότερα προγράμματα επελέγησαν φέτος από ό,τι είχε προγραμματιστεί στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών και ήθελα να μάθω γιατί. Συζητήσατε επίσης ε, για την απλούστευση των διαδικασιών και των, ε, εισγραφειοκρατίας. Ρωτώ λοιπόν σε ποιον ωφελεί η απλούστευση, όχι για τον πιθανό δικαιούχο. Αυτή την εντύπωση έχω σχηματίσει εγώ. Συζητώντας με διάφορους ανθρώπους του τομέα, διαμαρτύρονται έντονα ότι τα πράγματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, όλο και πιο γραφειοκρατικά και ότι αυτό αποτρέπει τους ανθρώπους από να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Μειώνεται το ενδιαφέρον τους. Τι προβλέπετε για να κάνετε τα πράγματα πραγματικά πιο φιλικά προς το χρήστη, πιο απλά. Γιατί ξέρετε, υποβαθμίζονται οι στόχοι μα όταν οι άνθρωποι διαμαρτύρονται σε τέτοιο βαθμό εξαιτία τη διαδικασία. Και μετά, όσον αφορά τα ε, προγράμματα μικρή κλίμακα που ε, αντιστοιχούν στο σκελετό του όλου θέματος. Πώς συμμετέχουν όλε οι χώρες ε, και πώς επιτυχάνεται η απαραίτητη ισορροπία. Τώρα για το κομμάτι των μέσων Ποιο είναι το ποσοστό μη επιλεξιμότητα των προγραμμάτων. Μπορείτε να μας πείτε κάποια νούμερα και μετά θέλω να πείτε πώς επιλέγετε τους εμπειρογνώμονες για τις επιτροπές για τα μέσα. Μιλήσατε για την εγγύηση δανείων που θα ξεκινήσει το 2016. Μπορείτε να μου πείτε πώς έχει προχωρήσει η επιλογή των οικονομικών διαμεσολαβητών και ποιος είναι επιφορτισμένος με αυτό, η DG e ή η DG ή e κάποια άλλη DG. Και μετά όσον αφορά την, την επικοινωνία, υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες και ιστότοποι των δύο γενικών διευθύνσεων. Δεν είναι πάντα συμπληρωματικές αυτές οι ιστοσελίδες, οι ιστότοποι και πολλές φορές είναι μόνο στα αγγλικά, το οποίο δεν βοηθάει ιδιαίτερα το χρήστη. Θέλω να σχολιάσετε παρακαλώ. Ευχαριστούμε. Έλγα για τις ε, πολύ ακριβείς σας ερωτήσεις. Ο κύριος Διακόνου θέλει να πει κάτι, δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να πει κάτι και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Ευχαριστώ. Έρχομαι σε αυτά που είπαμε και πριν για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά εγώ βέβαια στην αρχική μου τοποθέτησα, με τοποθέτηση προσπάθησα κάπως και να προκαλέσω. Βεβαίως και γνωρίζω ότι το σχέδιο είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια τελικά εσείς αποτελέσατε πρόκληση για μένα διότι κάθισα και προσπάθησα να τα σημειώσω όλα όσα είπατε και θα προσπαθήσω να περιλάβω στην εκθεσή μου. Τώρα επιτρέψτε μου να μου επιτρέψετε μάλλον εσείς οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθω σε επαφή και προσωπικά μαζί σας, να έρθω στα γραφεία σας, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες των όσων είπατε σήμερα. Ήταν ανακοίνωση υπηρεσία, όπω ε, την ονομάζουμε, να προσθέσω κι εγώ κάτι, γιατί δεν βλέπω να υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν να ρωτήσουν κάτι. Πρώτον, θα ήθελα να μου πείτε, όσον αφορά αυτό που είπατε προηγουμένω, για του διάφορου τομεί, ε, θέλω να σα ρωτήσω για τη σχέση μεταξύ τον προπολογισμό που έχουν προβλεφθεί κατά την άποψή σας αρχικά υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της πρόβλεψης των προπολογισμών και του ότι υπήρξε στα αιτήματα και το δεύτερο ερώτημα αφορά το ερώτημα της κυρίας Τρούπελ τις προϋποθέσεις επιλογής ενημερωθήκαμε αλλά καλά θα ήταν να το είχαμε επίσημα ενημερωθήκαμε ότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο εγκρίνει εμπειρογνώμονες ε, ομάδων η Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού και Παιδείας. Οι εμπειρογνώμονες που εγκρίνουν τα προγράμματα δεν είναι πια ομάδες, αλλά μεμονωμένα άτομα, online ουσιαστικά, ε, δύο άτομα νομίζω ε, συνιστούν τους εμπειρογνώμονες και κατά κάποιο τρόπο έτσι κάπως απομονωμένα κάνουν τη δουλειά τους. Το σύστημα αυτό κατά την αποψή σας ε, είναι πιο αποτελεσματικό ή μήπως τελικά είναι λίγο ε, γραφειοκρατικό λείπει ο διάλογος δηλαδή και για το νέο χρηματοδοτικό μέσο θα θέλαμε να καταλάβουμε θα θέλαμε να μάθουμε κατά πόσο υπήρξε κάποια δράση ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις εθνικές τράπεζες ώστε να συμμετάσχουν, ώστε να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια μεγάλη ευκαιρία. Και τέλος, στο πλαίσιο της Δημιουργικής Ευρώπης, έχουμε εντοπίσει κάτι που πρέπει να υλοποιήσει η Κομισιόν μέχρι το 2015, μια μελέτη επιπτώσεων για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Θέλουμε να μας πείτε σε ποια φάση βρίσκεται αυτή η μελέτη σκοπιμότητας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, δεν είπα παρακαλώ, έχετε το λόγο όποτε θέλετε. Thank you, Mrs. Chair. I will switch to English because I have papers with dates. Ευχαριστώ. Θα τα πω αγγλικά τώρα, επειδή έχω μπροστά μου κάποια έγγραφα με στοιχεία τα οποία είναι γραμμένα στα αγγλικά. Να ξεκινήσω δίνοντάς σας κάποια παραπάνω στοιχεία για τον αριθμό των σχεδίων που χρηματοδοτήσαμε το 2014, δηλαδή κατά τον πρώτο γύρο των ε, προκηρύξεων διαγωνισμών. Επικεντρωθήκαμε κυρίως ε, στο πρόγραμμα Culture και για το Media θα σας δώσω ε, στοιχεία, αλλά δεν είναι σαφές επειδή διαφέρει το σύστημα, δεν μπορώ να σας δώσω πολύ ξεκάθαρα στοιχεία. Για το πρόγραμμα πολιτισμός είναι τέσσερις συνιστώσεις προγράμματα συνεργασίας πρώτον. 411 συνολικά αιτήσει λάβαμε, μεγάλος αριθμός, εκ των οποίων χρηματοδοτήσαμε 58 σχέδια συνεργασίας, 21 μεγάλης κλίμακας και 37 μικρής κλίμακας. 40 εκατομμύρια ευρώ ήταν το συνολικό ποσό, λίγο πολύ. Λίγο λιγότερο από το προηγούμενο έτος, σας πενθυμίζω όμως ότι το πρόγραμμα είχε χαμηλότερο προπολογισμό το 2014 της Καμπύλης. Για τα προγράμματα λοιπόν συνεργασίας πιστεύουμε ότι έχουμε μια σχετικά ικανοποιητική ισορροπία σε ό,τι αφορά τους τομείς και τις χώρες. Εδώ έχω ένα στοιχείο που λέει ότι πάνω από 400 οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού συμμετέχουν στην διαδικασία επιλογής. Πολλοί δηλαδή. Δεύτερη συνιστόσα, δίκτυα για τα δίκτυα λάβαμε 58 αιτήσει και χρηματοδοτήσαμε 22 σχέδια. Συνολικός προπολογισμός περίπου 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα δίκτυα περιλάμβαναν 330 μέλη, άρα υπήρχε σημαντικό στοιχείο μόχλευσης ε, στη χρηματοδότηση αυτών των δικτύων. Η γεωγραφική κάλυψη δεν είναι βέβαια τόσο καλή όσο αυτή στα προγράμματα συνεργασίας. Έχουμε μεγάλο αριθμό δικτύων που προέρχονται από το Βέλγιο. Επειδή είναι πιο κοντά ε, στα θεσμικά όργανα τα δίκτυα για να παίρνουν πληροφορίες, ε, δημιουργεί αυτό μια συγκέντρωση και γι' αυτό το λόγο είχαμε πολλά από το Βέλγιο. Υπάρχει και μια συνέχεια με τα δίκτυα, άρα καλή ισορροπία νομίζω έχουμε. Σε ό,τι αφορά τη λογοτεχνική μετάφραση, 260 αιτήσει λάβαμε, επιλέξαμε 74 σχέδια. 3,5 εκατομμύρια το συνολικό ποσό πολύ ψηλότερο. 2,6 νομίζω ήταν το αντίστοιχο ποσό το 2013, άρα αισθητή αύξηση της χρηματοδότησης ε, των μεταφράσεων. Τέλος, πλατφόρμες, τέταρτη συνιστόσα. Η πιο καινοτόμος δεν υπήρχε στο πρόγραμμα πολιτισμός. Εκεί με τα χαράς είδαμε ότι είχαμε 24 αιτήσει. 5 από αυτές τις πλατφόρμες τις χρηματοδοτήσαμε 2,2 εκατομμύρια το ποσό. Και το ικανοποιητικό είναι μάλλον τα εξή δύο. Ότι είχαμε διαφορετικές προτάσεις ε, σε ό,τι αφορά τις χώρες, τους τομείς. 26 ε, μόνο χώρες εκπροσωπούνταν στις πλατφόρμες και οι αρμόδιοι κατάλαβαν τα βασικά. Τι είναι αυτά τα σχέδια, τι στόχο έχουν, ουσιαστικά να φέρουν κοντά τους καλλιτέχνες και να παραγάγουν καλά πολιτιστικά προϊόντα. Τα πήγαμε καλά. Θέλαμε να έχουμε και ένα νέο διαγωνισμό φέτο, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολλά υποσχόμενη αυτή η συνιστόσα. Για τα μίντια, ίσως η Λουθία να θέλει να πει κάποια. Εγώ ήμουν ο υπεύθυνο για τη διαχείριση του προγράμματο αυτού 2014. Δεν θα έχει αντίρρηση λοιπόν αν συνεχίσω. Ε, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αυτοματισμού, όπω είπα και πριν, στο μίντια. Έχουμε κάποια αυτόματα συστήματα διανομής και ανάπτυξης. Για τη διανομή, την ανάπτυξη, την πρόσβαση στις αγορές και τα φεστιβάλ, νομίζω ότι βλέπουμε να υπάρχει συνέχεια. Υπήρχαν όμως και κάποια νέα συστήματα στο media. Το πρώτο αφορά την ανάπτυξη του κοινού. Δεν ήταν και εξαιρετικά τα αποτελέσματα του πρώτου έτους, για να μην ειλικρινής, ίσως γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο το κόνσεπτ στις κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να βελτιώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές από φέτος. Δουλειά που έχει ήδη ξεκινήσει. Και για την επιγραμμική διανομή, το online distribution, δηλαδή νέες μορφές διανομής. Είχαμε ένα project το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, εξελόγηση συνεχίζεται και είχαμε και ένα νέο ε, για τα βιντεοπαιχνίδια για πρώτη φορά πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον του κλάδου. Φαίνεται δηλαδή ότι ενδιαφέρεται πολύ ο κλάδος αυτός για το πρόγραμμά μας. Τέλος. Τέλος, επαναλαμβάνω. Είχαμε, μάλλον χρειάστηκε να αναθεωρήσουμε το τι κάνουμε με το Europa Cinema, ένα ιστορικό εταίρο θα σας πω ποιες, μάλλον η Λουσία θα σας πει ποιες είναι οι προθέσεις για αυτό το δίκτυο, το πολύ μεγάλο δίκτυο. Σας ευχαριστώ. Πριν να μιλήσω για την ειδική αυτή περίπτωση, να σας πω λίγα γενικότερα νούμερα. Υπήρξε μεγάλος βαθμός συνέχειας σε αυτές τις διαδικασίες επιλογές για το πρόγραμμα των media. Λίγα ποσοστά για το 2014. Η εκπαίδευση έλαβε περίπου 7% του προϋπολογισμού που διαθέσαμε το 2014. Η ανάπτυξη 19, η παραγωγή και διεθνείς συμπαραγωγές περίπου 12%. Βλέπετε λοιπόν ότι το μεγάλο ποσοστό των χρημάτων πηγαίνει στην post-production, δηλαδή την προώθηση διανομή και πρόσβαση στις αγορές. Περίπου το μισό, 46% δηλαδή του συνολικού προπολογισμού πηγαίνει στη διανομή. Και νομίζουμε ότι η διανομή πάλι λαμβάνει εκεί, όπως είπα, μεγάλο ποσοστό. Το Europa Cinema και το Cinema Network είναι πολύ σημαντικοί δικαιούχοι, απολύπτες του προγράμματος. Έχουμε και τακτικές συζητήσεις κυρίως για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αυξημένη διανομή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών. Εκεί όπου υπάρχουν και λιγότερες κινηματογραφικές αίθουσες και επομένω η κυκλοφορία των ταινιών αυτών είναι και πιο δύσκολη. Γι' αυτό και αναζητούμε μαζί τους τρόπους να διανυμφθούν οι ταινίε αυτές και στις, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Νότιας Ευρώπης, όπου τα προβλήματα είναι περισσότερα. Αυτά. Θα σταματήσω εδώ. Ε, juste sur... Ε, ε, απλά να απαντήσω στις άλλες ερωτήσεις, η κυρία Τρέμπ ε, ρώτησε γιατί υπάρχουν λιγότερα προγράμματα συνεργασίας. Πολύ απλά, διότι ο προπολογισμό είναι μικρότερος και συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση που μπορούμε να δώσουμε στα συνεργατικά προγράμματα. Όπως είπα, είναι κάτι που τελειώνει το 2016. Το 2016 θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πολύ περισσότερα προγράμματα επικοινωνίας. Η κυρία Τρίπελ ε, υπενθύμησε επίσης ότι η διαχείριση του προγράμματος δεν είναι και οι απλούστεροι και ούτε οι, πιο, οι δημοκρατικότεροι δυστυχώ πρέπει να, συμφωνήσω μαζί σα. Οι προσπάθειε απλούστευσης δυστυχώ, δεν απέφεραν αποτελέσματα ειδικότερα η χρήση των ηλεκτρονικών αιτήσεων ε, και εντύπων δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί πλήρω. Επίση χρησιμοποιήσαμε αποκοπή ποσά μόνο σε ορισμένε περιπτώσει και δεν έχουμε λάβει feedback. Και εγώ λυπάμαι που δεν καταφέραμε να απλουστεύσουμε περισσότερο τη διαχείριση του προγράμματος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι είναι συνέπεια μιας προσπάθειας διασφάλισης ε, τη χρηστής διαχείριση αυτού του προγράμματος. Δεν ξέρω πώς να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, Αν απλουστεύσουμε τη διαχείριση του προγράμματος εκτεθέμεθα σε ένα κίνδυνο πική διαχείριση. Και ίσω μερικέ φορέ ε, υπερβάλλουμε ε, έχοντα αυτή τη, μέρημνα, τη διαρκή μέρημνα για την ασφάλεια. Έχω απόλυτη συνείδηση των όσων είπατε. Όμω, όσον αφορά του ιστότοπου, γίνεται προσπάθεια προσέγγιση των ιστοτοπών που αφορούν το πρόγραμμα και εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε με τον οργανισμό μεταξύ οργανισμών ώστε να συγκλίνουν οι ιστότοποι Συνεργαζόμαστε και με την DG Connect ώστε τα δύο υποπρογράμματα να αποτελέσουν το αντικείμενο κάποιε. Ε, να, να επικοινωνούν σωστά μεταξύ του. Για το ζήτημα των εμπειρογνωμόνων, ε, αν μου το επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα δώσω το λόγο στον, κύριο, στον συνάδελφο μου τον Καρλ Μπαρτάκ. Τώρα για τα χρηματοδοτικά μέσα και τις κεντρικές τράπεζες θα απαντήσει η συναδελφός μου. Γεια σας, καλησπέρα. Όπως γνωρίζετε, η επιλογή, η αξιολόγηση όλων των αιτήσεων στο πλαίσιο του Δημιουργική Ευρώπη πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της εκτελεστικού οργανισμού και της Επιτροπής από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Το σύστημα έχει αλλάξει σε σχέση με το τελευταίο πρόγραμμα, διότι για τα περισσότερα προγράμματα λειτουργούμε εξ αποστάσεως. Δεν καλούμε πλέον τους εμπειρογνώμονες να έλθουν στις Βρυξέλλες και να καθίσουν μαζί μας και να συνεργαστούμε για τα προγράμματα. Το κάθε πρόγραμμα αξιολογείται από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες που επιλέγονται ανάλογα με τις ικανότητές τους και εγκρινούν το πρόγραμμα με αμοιβαία συνεργασία και όταν καταλήξουν σε συνένεση ε, βάσει κάποιων κριτηρίων ε, και κάποιων βαθμών εγκρίνεται το πρόγραμμα. Όταν υπάρχει σημαντική διχογνωμία μεταξύ των δύο εμπειρογνωμόνων επί 30 περισσότερων σημείων, τότε καλείται ένα τρίτο εμπειρογνώμων να, να παρέμβει και σε αυτός ο τρίτο εμπειρογνώμων προτείνει κάποια συνένεση και αν επιτευχθεί αυτή η συνένεση και από τους τρεις τότε ο, ο βαθμός αυτός πόντων αποδίδεται στο πρόγραμμα. Πέραν αυτού Βάσει των διδαγμάτων που αποκομίστηκαν το 2014 για το 2015 θα ξεκινήσουμε να συνεργαζόμαστε με μια ομάδα ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων που θα αξιολογούν τα προγράμματα εκείνα τα οποία είναι οριακά ανάλογα δηλαδή με τα χρήματα που υπάρχουν διαθέσιμα κάποια στιγμή πρέπει να πούμε θα επιλέξουμε αυτό τον αριθμό προγραμματών συνεργασίας αυτή είναι η διαχωριστική γραμμή αυτό είναι το όριο 18 για παράδειγμα πόντων ή 80 πόντι και θα πούμε ότι υπάρχει κάποια γκρίζα ζώνη δηλαδή πόντων ουσιαστικά. Τα προγράμματα που βρίσκονται λοιπόν σε αυτή την γκρίζα ζώνη θα επαναξιολογούνται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες του εκάστοτε προγράμματος, θα λαμβάνουν επίσης υπόψη τη γεωγραφική ισορροπία, θα λαμβάνουν υπόψη την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων υποτομέων, και η πρότασή τους μετά θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Επιλογής. Η τελική απόφαση λαμβάνεται πάντα από την Επιτροπή Επιλογής η οποία αποτελείται από αξιωματούχους της Επιτροπής και του εκτελεστικού οργανισμού. Ελπίζω να σας εξήγησα κάπως καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε από το 2015. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα θα ήθελα να απαντήσω σε δύο πρόσθετα ερωτήματα, ετσι πάνω στα ερωτήματα τα οποία αφορούσαν το ένα, αυτό που είπε η κυρία Τρούπελ για τα φεστιβάλ, τη μη επιλεξιμότητα φεστιβάλ. Ο αριθμό των προτάσεων που λάβαμε για φεστιβάλ ήταν πάρα πολύ ψηλό. 316 συγκεκριμένα από 33 χώρες. Από όλα αυτά επιλέξαμε 88 φεστιβάλ από 25 χώρες και αυτά τα επιλέγοντα φεστιβάλ νομίζω ότι πρόσφεραν μια ισορροπία. Δηλαδή είχαμε παγκόσμια φεστιβάλ, νεανικά φεστιβάλ, φεστιβάλ ε, ταινιών μικρού μήκους κτλ. Τι έγινε λοιπόν φέτος, η ποιότητα των προτάσεων ε, δεν ήταν καθόλου ομοιόμορφη, είχαμε πολύ υψηλή πρόταση και πολύ χαμηλής ποιότητα προτάσεις και θέλαμε τα ε, σχέδια που θα επιλέξουμε να έχουν πολύ στενοβούς μηχανισμούς ανάπτυξης κοινού. Audience development, όπως το λέμε. Ίσως σε κάποιες ε, περιπτώσεις δεν δόθηκε ιδέωσα προσοχή σε αυτό το πολύ σημαντικό όμως, κατά εμάς, κριτήριο. Κυρία Τρύπρη, πόσα φεστιβάλ επιλέξατε? 88 είναι η απάντηση, από 25 χώρες. Τώρα, στο ερώτημα της κυρίας Κώστα για την επιλογή των ε, ενδιάμεσων δικαιούχων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, ε, με βάση τη συμφωνία εκχώρηση αμμουδετών, θα πάρει την απόφαση. Οι παράμετροι όμω αυτή τη άσκηση, αυτού του εγχειρήματο, ορίζονται από την νομική βάση του προγράμματο Δημιουργική Ευρώπη. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων είναι ε, το εκτελεστικό όργανο, ο εκτελεστικός φορέας, αλλά θα λάβει πλήρω υπόψη τα κριτήρια της νομική βάσης που περιλαμβάνονται στην ε, συμφωνία συνεργασίας που συνάπτουμε με το ΑΕΦ. Πρόεδρος, αν με επιτρέπετε να θέσω δύο συμπληρωματικά ερωτήματα. Για τον υποτιτλισμό, είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπαμε εμείς υποτιτλισμός και μεταγλώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσον λάβατε κάποια αιτήματα ήδη. Νομίζω ότι υπήρχε ένα πιλωτικό σχέδιο με το παράδειγμα του βραβείου Λουξ. Και οι σχέσεις με τις τρίτες χώρες είναι ένα άλλο θέμα που με απασχολεί. Δεν έχουμε το Media Mundus, αλλά έχουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με τρίτες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσο έχετε συνάψει ήδη κάποια συμφωνία ή αν σε παλαιότερες συμφωνίες προστίθεται συγκεκριμένο σκέλος. Δεν ξέρω κατά πόσο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το θέμα. Πού βρισκόμαστε τέλος πάντων. Ναι, πράγματι υπάρχουν ευκαιρίες ε, συνεργασίας με τρίτες χώρες. Και τα Ταμεία Διεθνών Συμπραγωγών ε, είναι παράδειγμα των συνεργασιών που σκόπευαμε να αναπτύξουμε με τρίτες χώρες. Προσπαθώ τώρα να βρω, ε, για να σας δώσω πληροφορίες για την εκπαίδευση στα φεστιβάλ και αυτή είναι ένα παράδειγμα. Προσπαθώ να βρω προφορίε για τα ταμεία διεθνού συμπαραγωγής που έχουν επιλεγεί. Προσπαθώ να βρω προφορίε. για αυτό. Perhaps, Να σα ε, δώσω μια γενική εικόνα όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Όπω γνωρίζετε η νομική βάση προβλέπει τη συμμετοχή χωρών εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε ανοίξει ευθύ εξ αρχή το πρόγραμμα, ανέκαθεν το πρόγραμμα αυτό στι τρίτε χώρε και από την αρχή είχαμε τη συμμετοχή των χωρών τη ΕΖΕΣ όπως και στα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα. Επίσης έχουμε συμμετοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των υποψήφιων χωρών και θα υπάρχουν και υποψήφιες χώρες από τα Βαλκάνια. Οι δύο μόνες εξαιρεσει είναι η Ελβετία αφενός λόγω των γνωστών αιτιών. Όλα σταμάτησαν με την Ελβετία. Με την Ελβετία διαπραγματευόμαστε, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε το πρόγραμμα για αυτούς και έχουμε και κάποια καθυστέρηση με την Τουρκία. Ενώ, καθυστέρηση ενός έτους ε, για οικονομικούς ε, λόγους, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2015 συμμετέχει η Τουρκία. Οι χώρες αυτές ε, οι περισσότερες συμμετέχουν και στο υποπρόγραμμα πολιτισμού, αλλά όχι στο υποπρόγραμμα μέσων, διότι δεν έχουν ευθυγραμμίσει την νομοθεσία τους με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία περί οπτικοακουστικών υπηρεσιών, που αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή στο υποπρόγραμμα για τα μέσα. Πέραν αυτού, έχουν υπάρξει αιτήσει από τρεις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας και έχουμε οριστικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία. Αυτές οι τρεις χώρες λοιπόν θα συμμετάσχουν στο υποπρόγραμμα πολιτισμού ήδη από το 2015. Επίσης ε, έχουμε και ε, επιθυμίες συμμετοχής από κάποιες χώρες της νότιας γειτονίας αλλά δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Για να επανέλθω στο ζήτημα των πιθανών συνεργασιών με τρίτες χώρες. Πρώτον λοιπόν με το τα Ταμεία Διεθνών Συμπαραγωγής αφορούν, είναι κονδύλια που αφορούν τις συμπαραγωγές με τρίτες χώρες. Πέντε ταμεία ε, έχουν επιλεγεί και θα αρχίσουν να υλοποιούν τις ε, δραστηριότητές τους φέτος. Αυτό είναι το ένα. Μετά η ενσωμάτωση του Media Mundos ε, έχει γίνει μέσω της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στην αγορά. Στο κομμάτι της εκπαίδευσης τα αποτελέσματα ήταν κάπως απογοητευτικά λόγω του περιορισμένου αριθμού των δικαιούχων. Ουσιαστικά είναι μόνο τέσσερις. Για το κομμάτι της πρόσβασης στην αγορά, η ενσωμάτωση του μου ιδιαμούντος ε, οδήγησε σε αυξημένο επίπεδο αιτήσεων και ζήτησης αλλά τα προηγούμενα προγράμματα του Μόντους πρέπει να ξέρετε δεν ε, απέδωσαν πολύ καλά σε αυτό το γύρο. Συνεπώς είναι περιορισμένος ο αριθμός προγραμμάτων που ενσωματώνονται στο νέο πλαίσιο. Τέλος, να πω ότι όσον αφορά τον υποτιτλισμό, είναι πλήρες επιλέξιμο κόστος υπό το μηχανισμό διανομής γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και εντάσσεται πλήρως στο μηχανισμό διανομής. Ε, e Αναμένω ακόμα μια απάντηση, δεν ξέρω αν και άλλοι συνάδελφοι έχουν ικανοποιηθεί. Σας ευχαριστώ για όλα σε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες. Για τους δείκτες, δεν μου είπατε, τους δείκτες πολιτισμού, τους πολιτιστικούς δείκτες που για μας είναι πολύ σημαντικοί. και για τη μελέτη σκοπιμότητας. Ξέρουμε ότι έγινε μια πρόσκληση από την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού. Θέλω να μου πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει ήδη η δουλειά. Δεν είναι κάτι απλό. Θα το θυμάστε κι εσείς κυρία Πρόεδρε. Πάντω σίγουρα πρέπει να έλθει σε αίσιο πέρα. για να ολοκληρώσουμε και την ε, αξιολόγηση του 16-17, άρα συνεχίζεται. Η Λουθία. Θέλω να προσθέσω ότι στους δείκτες αυτούς θέλουμε να συνεργαστούμε από κοινού, να, στενά μάλλον, γιατί αφορά τον πολιτιστικό δημιουργικό κλάδο και εκεί πρέπει να γίνει ακόμη η δουλειά. Χέρι με χέρι προχωρούμε από κοινού οι διευθυντικές διευθύνσεις για αυτούς τους δείκτες. Ευχαριστούμε. Εγώ αναφέρθηκα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο όμως ε, αφορούσε τη μελέτη σκοπιμότητας που θα παρουσιαστεί νομίζω όμως τον Ιούνιο του 2015 και προβλέπει αν δεν απατώμε κάτι διαφορετικό από τα όσα έχουν γίνει ήδη από το παρατηρητήριο οπτικοακουστικών μέσων. Είναι μια άλλη πτυχή που αφορά τους δείκτες των πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων και που αφορά την Γενική Διεύθυνση Πολιτισμού. Ήθελα απλά να μου διαβεβαιώσετε ότι η προθεσμία είναι τον Ιούνιο του 2015. Euh, oui, me dit que ce sera effectivement prêt. Ναι, μου λένε ότι θα είναι όντω έτοιμη για τον Ιούνιο του 2015. Εξαιρετική. Εξαιρετικό νέο. Μας χαροποιεί ιδιαίτερος. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Το κύριε Μανιά και του συναδέλφου του. Σας ευχαριστούμε για την ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Η ενημέρωση αυτά για μας ήταν πολύ ωφέλιμη και σημαντική και η εμβάθυνση των διαφορών θεμάτων και ο κύριος Επιτρόπος μας κάλεσε για μια κοινή επίσκεψη στον οργανισμό σας ε, ώστε πιο άμεσα να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το πρόγραμμα αυτό που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Εφάγομαστε λοιπόν ε, το έργο των δύο Γενικών Διευθύνσεων ένα αποτελεσματικό χωρίς κατακαιρματισμό του προγράμματος. Ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για αυτή την μεγάλη συνεδρίαση. Είμαστε εδώ από χθες το απόγευμα. Ευχαριστώ τη Γραμματεία που μας στήριξε και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη συνεδρίαση αλλά και πριν από αυτή στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας.